Ε, good afternoon, everybody. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τώρα έχω στη διάθεσή μου ό,τι χρειάζομαι για να κηρύξω την έναρξη της συνεδριάσεως. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ας αρχίσουμε την συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής ΛΥΜΠΑ. Έχουμε τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πρώτα απ' όλα έχουμε την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα σε ποινικέ υποθέσεις με εισηγητή τον κύριο Μέλου. Στη συνέχεια έχουμε την κατάσταση στην Ουγγαρία, τη παρουσία του κύριου Ντεβάλ που είναι ο Γενικός Διευθυντής Δικαιοσύνης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ω τελευταίο σημείο έχουμε το πολιτέ πλαίσιο για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2013 2017. Ως καθώς μάλλον ο πρόεδρος της Επιτροπής μας δεν είναι εδώ σήμερα το απόγευμα, αναλαμβάνω εγώ να προεδρεύσω για αυτό το απόγευμα. Να γνωρίζετε όμως ως Ουγγαρέζα, μέλος της Επιτροπής αυτής και ως ε, απλό μέλος αυτής της Επιτροπής, θα ήθελα να πάρω το λόγο στο επόμενο θέμα. Οπότε θα ζητήσω στη Σόφη να προεδρεύσει για λίγο, αν δεν έχετε και εσείς πρόβλημα με αυτό, για να μπορέσω κι εγώ να μιλήσω υπό την ποιότητα του μέλους της Επιτροπής αυτής. Πρώτο θέμα, λοιπόν, είπαμε, είναι η έκδοση οδηγίας ε, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα σε ποινικέ υποθέσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα τη αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών μέτρων γιατί εμπλέκονται διαφορετικά συνταγματικά συστήματα και διαφορετικές ε, προδιαγραφές. Είχαμε ήδη εξετάσει από πέρυσι το θέμα αυτό. Σήμερα έχουμε εδώ τον κύριο Μέλο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών θα είναι Ιανουαρίου το απόγευμα στις 5. Παρακαλώ κύριε Μέλο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό είναι όντως πολύ σημαντικό, αλλά και αρκετά επίμαχο. Ξέρετε ότι ο βασικός μας στόχος είναι η ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων και αγαθών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως τίθεται και θέμα κυριαρχίας πρώτα απ' όλα των χωρών μελών. Οι αστυνομικές αρχές, οι αστυνομικοί γενικά δεν μπορούν να πάνε από τη μία χώρα στην άλλη, να περάσουν στα σύνορα δηλαδή για να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά τους. Όμως θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη αποτελεί ένα χώρο δικαιοσύνης και ότι η ελευθερία κυκλοφορία ατόμων και αγαθών δεν σημαίνει από την άλλη μεριά αύξηση της εγκληματικότητα. Συνεπώς, η πρώτη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας με την πρωτοβουλία αυτή είναι από τη μια να φροντίσουμε να ερευνάται η εγκληματικότητα σωστά παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη μεριά, συγχρόνως δηλαδή, να μην υπονομεύσουμε την δικαιοσύνη και τα κυρίαρχα δικαιώματα των κρατών μελών. Να μην αφισβητούμε δηλαδή τις συνταγματικές ή νομικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ χωρών μελών. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με τις τροπολογίες μου ελπίζω να έχω καλύψει πολλές από τις ανησυχίες των συναδέρφων. Πολλά, πολλοί συνάδελφοι μάλλον, συμφώνησαν για διάφορα σημεία και πολλοί συνάδελφοι επίσης έκαναν ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχω συμπεριλάβει όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές. Ε, κάποιοι συνάδελφοι εξέφρασαν ανησυχίες όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής. Νομίζω ότι τους κάλυψα. Και για όσου δεν έχουν διαβάσει ακόμα την έκθεσή μου αυτή, θα σας πω ποια είναι τα κύρια σημεία της. Βασιζόμαστε σε απόφαση αρμόδιων ε, νομικών αρχών των κρατών μελών. Η ιδέα δηλαδή είναι να επιτρέψουμε ε, έρευνα για εγκληματικούς λόγους να γίνεται ε, σε μία χώρα μέλος εφόσον την έχει ζητήσει κάποιο άλλο. Αυτό είναι το θέμα της αμοιβαία αναγνώρισης. Προσπάθησα, δεν ξέρω αν τα κατάφερα, αλλά τουλάχιστον προσπάθησα να διασφαλίσω ότι η εφαρμογή αυτής της αρχής της αμοιβαία αναγνώρισης δηλαδή δεν αντιβαίνει και δεν θίγει συνταγματικά ε, δικαιώματα. Δεν έρχεται δηλαδή σε αντίθεση με συνταγματικές προδιαγραφές ή νομικές προδιαγραφές που ισχύουν στις διάφορες χώρες. Νομίζω ότι καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τα επίμαχα σημεία. Αστυνομικές αρχές που ζητούν να γίνουν έρευνες σε άλλη χώρα μέλος ή ζητούν συλλογή στοιχείων, αποδεικτικών στοιχείων κτλ. Δεν μπορούν να το κάνουν χωρίς να υπάρξει παρέμβαση κάποιου νομικού ή δικαστικού σώματος. Βέβαια μπορούν και να αρνηθούν προκειμένου να αποφύγουν παραβίαση του συντάγματός τους κάποιες χώρες ή άλλες νομικές προδιαγραφές που ισχύουν. Να αποφύγουν παραβίαση αυτών των προδιαγραφών. Για παράδειγμα, πάνω πάνω στον κατάλογο αυτών των περιπτώσεων έχουμε την αρχή της διτής ε, δίκης. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να δικαστεί δύο φορές για το ίδιο αδίκημα. Αυτή είναι μια αρχή την οποία διασφαλίζουμε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός είναι ένας λόγος άρνησης αιτήματο έρευνας. Δεύτερον, δεν υπάρχει υποχρέωση να δώσει συνέχεια μια χώρα εφόσον ένα δίκημα σε μια χώρα δεν είναι δίκημα και στην άλλη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η άλλη χώρα, η δεύτερη χώρα, μπορεί, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να προχωρήσει σε έρευνα. Έπειτα υπάρχει και το θέμα της εδαφικότητας, γιατί εδώ πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι, ότι το έγκλημα έχει λάβει χώρα στο κράτος Α, ώστε να τηρείται ώστε να τηρούνται να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα και των δύο χωρών. Δηλαδή είναι θέμα σεβασμού των δικαιοδοσιών των δύο χωρών. Ε, γι' αυτό και εδώ δέχτηκα την πρόταση που μου έκαναν συνάδελφοι, ιδιαίτερα από την Βόρεια Ευρώπη, σχετικά με το θέμα αυτό της δικαιοδοσίας. τίποτε περιορίζει την ελευθερία έκφρασης ή την ελευθερία τύπου ε, υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία όπου αυτοί οι κανόνες είναι πολύ συγκεκριμένοι και ακριβώς γι' αυτό βάλαμε αυτήν εδώ την διατύπωση. Ή επίσης όταν ε, γίνεται παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αυτά προβλέπονται στο συγκεκριμένο χάρτη ή στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή όταν θεωρείται ότι ένας δικαστής δεν επικύρωσε το μέτρο και Υπάρχουν, ε, δίνω και κάποια παραδείγματα και θα, και έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε ολόκληρη την πρόταση. ώστε να είναι βέβαιη η επιβολή του νόμου και η, στην δικαιοδοσία του κάθε κράτους. Και θα ήθελα να πω ότι θεσπίζονται προθεσμίες ώστε το, γιατί το δίκαιο άνευ προθεσμιών μπορεί να είναι τελικά άνευ ουσίας και μπορεί κάποια υπόθεση να ζημιωθεί αν δεν δοθούν οι απαραίτητες αποδείξεις στις κατάλληλες προθοσμίες που να είναι πάντως λογικές. Όλοι μας γνωρίζουμε παραδείγματα διασυνοριακής εγκληματικότητας όπου λόγω έλλειψης πλήρωσης των προθεσμιών ε, πέρα ας πούμε από την, ε, το Eurojust ή ποινική διαδικασία ζημιώνεται. Γι' αυτό και λέμε ότι θα πρέπει να γίνεται η εκτέλεση όσο γίνεται πιο σύντομα, μέσα σε μια προθεσμία 30 ημερών μετά από το αίτημα. Ωστόσο, το κράτος που λαμβάνει το αίτημα μπορεί να ζητήσει μια παράταση της προθεσμίας εφόσον υπάρχει αιτιολογημένο το αίτημα. Αυτά, Πρόεδρε. Έχω κάθε ενδιαφέρον να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων από, τα διάφορες, από τις διάφορες ομάδες, τους και ηγητές, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, έτσι ώστε το τέλος να έχουμε ένα καλό σχέδιο που γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την έρευνα σχετικά με τα δικήματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μέλο. Πριν να στραφώ στους συναδέλφους και να αρχίσει η συζήτηση, θα ρωτήσω το Συμβούλιο και την Κομισιόν αν θέλουν να παρέμβουν. Το Συμβούλιο. Μάλιστα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως αναφέρατε, το Συμβούλιο έφτασε σε μια γενική προσέγγιση για αυτό το θέμα στην ε, διαβούλευσή του το Δεκέμβριο και προσβλέπουμε στην έναρξη των διαπραγματεύσεων για αυτή την υπόθεση. Μόλις λάβαμε βέβαια το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή εχθές, αλλά εκ πρώτης όψεως είμαστε πολύ ε, θετικοί. Βλέπουμε ότι η έκθεση συμπεριλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που αντιστοιχούν στις ε, διαβουλεύσεις που κάναμε και στο Συμβούλιο όπως για παράδειγμα η ένταξη της ε, δοκιμής ε, αναλογίας καθώς και η απέτηση από το κράτος έκδοσης ε, του εντάλματος έρευνας και του κατά πόσο αυτό είναι απαραίτητο και αυτό συζητήθηκε και συμπεριλήφθηκε στη γενική προσέγγιση στην οποία συμφωνήσαμε το Δεκέμβριο. Επίσης, πρόταση ε, για να μπορούμε να εξασφαλίζουμε την πρόσβαση στις ε, νομικές ε, αποφάσεις. Ίσως βέβαια σε κάποια άλλα σημεία θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο. Η συγκητής ανέφερε τώρα στην ομιλία του το θέμα της εμπλοκής των δικαστικών αρχών. Αυτός είναι ένας τομέας όπου θα χρειαστεί να εργαστούμε περισσότερο. Και επίσης επιπλέον βάση για την άρνηση όπως ε, για παράδειγμα το διπλό, ε, η διπλή επιβολή ποινής. Πάντως καλωσορίζουμε το σχέδιο έκθεσης και προσβλέπουμε στην συνεργασία και στις διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και στρέφομαι στην Επιτροπή. Θα θέλατε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μέλο, τον εισηγητή, και να πω ότι όπως και η Προεδρία Χαιρόμαστε για αυτή την έκθεση που θεωρούμε πως αποτελεί εξαίρετη βάση για συζήτηση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για τη συναπόφαση. Η ε, Κομισιόν συμμερίζεται την άποψη του κυρίου Μέλο ε, για το ότι είναι απαραίτητο το μέτρο του, Ευρωπαϊκού Εντάλματος Ερεύνης για την έρευνα σε ποινικό ε, χώρο και συμβάλλει στη δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης για να απαντήσουμε, να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της σημερινής ε, πραγματικότητας και να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Αυτός ο χώρος δικαιοσύνης βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην αρχή αμοιβαία αναγνώρισης που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δικαστική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η διευκόλυνση της ε, απόκτησης αποδείξεων όπως ε, αποπειράται να κάνει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερεύνης θα συμβάλλει στην σωστή εξέλιξη της ποινική διαδικασίας. Είναι σαφές ότι οι δικαστές εισαγγελείς στην Ευρώπη σήμερα χρειάζεται να συνεργάζονται όλο ένα και πιο στενά για να προστατέψουν τους πολίτες και για να αποκαταστήσουν τα δικαιώματα των θυμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι για να είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό και σύγχρονο αυτό το μέσο του εντάλματος έρευνας και η δικαστική συνεργασία και να τηρούνται οι λογικές προθεσμίες που ανέφερε ο εισηγητής, αυτή η συνεργασία θα πρέπει να είναι ε, ε, ρευστή, να ρέει δηλαδή όσο γίνεται περισσότερο και το ένταλμα να αποτελεί πρόοδο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς αλληλοβοήθειας, αρρωγής, που βασίζεται στην καλή βούληση, στην καλή θέληση των κυρίαρχων κρατών να συνεργαστούν ή όχι αναπερίπτωση. Αυτό σημαίνει βέβαιως ε, εμπιστοσύνη ανάμεσα σε κράτη που έχουν κοινέ αξίες δικαστικές, ε, τήρηση και σεβασμό των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων Σημαίνει επίσης πως το ένταλμα ερεύνης θα πρέπει να αναγνωρίζεται από τα κράτη-μέλη με τις λιγότερες ε, δυνατές διατυπώσεις, χωρίς ε, να ζημιώνεται βεβαίως το θεμελιώδες δικαίωμα του τεκμηρίου ε, αθωότητας. Προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα σύγχρονης έρευνας στο κεφάλαιο 4, όπως για παράδειγμα οι πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η Κομισιόν τέλος να πω ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του εισηγητή για τη σημασία που αποδίδει στον σεβασμό των διαδικαστικών ε, δικαιωμάτων των ατόμων που είναι υποπτά μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Ερεύνης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι όλα τα μέτρα για το, σε σχέση με τον οδηγό και κυρίως η οδηγία για την πρόσβαση σε ε, δικηγόρο στόχο έχουν να ασφαλίσουν το πλαίσιο των διαδικαστικών δικαιωμάτων μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται και το αίτημα για ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνας. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί καλή ισορροπία μέσα σε αυτό το κείμενο που είναι πολύ σημαντικό για τον κοινό ε, χώρο δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ και στρέφομαι στους συναδέλφους. Μπορείτε να πάρετε το λόγο. Έχω έξι ονόματα στον κατάλογό μου. Mr. Πρώτος ο κύριος Κροτσέτα. Σας ευχαριστώ. Εγώ είδα πως η έκθεση του συναδέλφου Μέλο εισάγει κάποια ερωτήματα αλλά ε, και είδα μάλιστα ότι και εγώ ως εκπρόσωπος της ομάδας των σοσιαλιστών αλλά και ο συνάλφος Άλμπρεχτ και άλλοι είχαμε θέσει κάποιες εγγυήσεις όσον αφορά, είχαμε ζητήσει μάλλον κάποιες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και αυτή η πτυχή είναι πολύ σημαντική. Η δική μας αξιολόγηση όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα ε, έρευνα είναι, κάτι το, είναι, είναι κάτι το απαραίτητο και ε, θεωρώ πως το Συμβούλιο καλά έκανε να προτείνει αυτή την πρωτοβουλία. Είναι προφανές ότι πολλά αδικήματα ή και εγκλήματα κάποιες φορές δεν μπορούν να διωχθούν γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικέ δυνάμεις ή τις εισαγγελίες των διαφόρων χωρών. Άρα λοιπόν προκύπτει ε, κάτι το τελείως νέο από δικαστικής άποψης όπως έλεγε ο συνάδελφος Μέλο που βασίζεται στην αμοιβαιότητα αναγνώρισης με την έννοια ότι κάθε χώρα αναγνωρίζει ότι η άλλη έχει κάνει το σωστό. Αυτή η αξιολόγηση θεώρησα ωστόσο από την αρχή ότι είναι υπερβολική. Διότι η αξιολόγηση της ίδιας της λογικής στο έγγραφο του Συμβουλίου δεν εγγυάται τον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών. και τα θεμελιώδη δικαιώματα, γιατί γνωρίζουμε ότι όλες οι νομοθεσίες σε όλα τα κράτη-μέλη δεν είναι πάντα ομοιογενείς. Αν αφήσουμε κατά μέρος τον τύπο, την ελευθεροτυπία, αλλά ας πούμε, τα, όσα τα, τα ρεπορτάζ μας φτάνουν από την Ουγγαρία ε, θέτουν ε, προβλήματα για την ευρωπαϊκή συνείδηση σε ένα βαθμό πολύ ε, υψηλό και γι' αυτό ας πούμε θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με ένα ένταλμα ερεύνης που ξεκινάει από την Ουγγαρία που ανοιχτά παραβιάζει το κοινοτικό δικαίωμα, τα δικαιώματα των διαφόρων κρατών αλλά και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης. Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα και ο Μέλο έχει εδώ εισάγει διάφορα στάδια, όμως υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει καλύτερα να διευκρινιστούν και να ενισχυθούν. Για παράδειγμα, έχουμε επιτέλους, και αυτό είναι κάτι που Εξ αρχής το ζητήσαμε το ένταλμα να εκδίδεται από έναν οργανισμό που να είναι δικαστικός. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ένας οποιοδήποτε αστυνομικό ή μια οποιασδήποτε χώρας που ζητά από τον αστυνομικό μιας άλλης χώρας κάτι χωρίς αυτό να επικυρωθεί από οποιοδήποτε εισαγγελέα να κάνει μια έρευνα γιατί αυτό θα ήταν επιστροφή στο κράτος το αστυνομικό. Ε, δεν θα ήταν δικαστική συνεργασία και δεν θα συμφωνούσε με τις βασικές ευρωπαϊκές αρχές. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ένας εισαγγελέα που εξ αρχής το επικυρώνει αυτό το ένταλμα. Αλλά υπάρχει και το εξή πρόβλημα. Ποιος εκτελεί το ένταλμα, γιατί πριν έλεγε ο μέλος αν είναι ένας ε, ε, ε, κάτι παράνομο που έχει γίνει σε μια συγκεκριμένη χώρα. Εντάξει, αλλά ποιος θα εκτιμά αυτό. Μια οποιαδήποτε αρχή που επικυρώνεται από τις διεθνείς αρχές. Όχι. Σύμφωνα με το κράτος δικαίου και σύμφωνα με τις αρχές της ελευθερίας που διέπουν την Ευρώπη, ένας εισαγγελέα θα πρέπει να κρίνει κατά πόσο είναι νόμιμο ή παράνομο ένα πράγμα. Δεν μπορεί να είναι άλλη αρχή που το εκτιμά αυτό, γιατί θα μπορούσε να είναι κάτι τελώς παράνομο, ακόμα και από πλευράς των πολιτικών αρχών ε, ενός αδικήματος. Γι' αυτό και πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ποια είναι τα δικαιώματα των ε, διαδίκων και θα πρέπει αυτά να γίνουν σεβαστά. Έπειτα, σε ποιον θα πρέπει να αντιταχθεί ο διάδικος. Ο κατηγορούμενος, ας πούμε, ο Ούγγρος, ο Ιταλός ή ο Άγγλος. Αν είναι Ιταλός, ας πούμε, πρέπει να περάσει δίκη στην Αγγλία ή στην Ουγγαρία, θα είναι πολύ δύσκολη η υπόθεση. αγγλια η στην ουγγαρια θα ειναι πολυ δυσκολη υποθεση γιατι Μπορεί να μιλάμε για το δικαίωμα στην νομική αρρωγή κτλ. ή ό,τι θέλουμε, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο πολίτης να βρίσκεται σε μια ισότιμη θέση. Εγώ μάλιστα είμαι μεταξύ άλλων όπου σε πολύ σοβαρά δικήματα είστε στο οργανωμένο έγκλημα, θα τους έκλεινα μέσα και θα πέταγα στο πηγάδι τα κλειδιά. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να ενεργούμε έτσι. Ε, τα δικαιώματα των πολιτών είναι απαραβίαστα και άρα ορισμένα ορόσημα θα πρέπει να τεθούν έτσι ώστε να ενισχυθεί το κείμενο γιατί θέλουμε τη μέγιστη δυνατή συνεργασία όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας. Χαιρετίζουμε θετικά την πρωτοβουλία του Συμβουλίου γιατί τη θεωρούμε σημαντική. Αναγνωρίζουμε πω ο εισηγητή έκανε σπουδαία δουλειά, αλλά ότι ορισμένα ζητήματα που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα θα χρειαστεί να αποτελέσουν μέρος αυτή της έκθεση. Ευχαριστούμε, ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω γερμανικά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Μέλο. Η έκθεσή του είναι όντως ένα καλό πρώτο βήμα, πολύ σημαντικό και καλό είναι που μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα, διότι το Συμβούλιο προσπαθεί να συμφωνήσει και πρέπει να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση και να πούμε στο Συμβούλιο ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε. Κατά δεύτερον λόγο πρέπει να σας πω ότι θεωρώ πολύ καλό ότι τα θέματα που αναφέρθηκαν για τη σχετικότητα των αρχών Νέμπες και Ίντεμ και του τομέα της εδαφικότητος λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή θεωρώ ότι αυτό το σχέδιο είναι πολύ καλό. Έχω να κάνω και ορισμένες περαιτέρω παρατηρήσεις, διότι ο κύριος Κροτσέτα είπε τώρα ότι ιδιαιτέρως στο θέμα της αναλογικότητος και στα θεμελιώδη δικαιώματα δεν χρειάζεται να προβούμε σε μία προσθήκη και μάλλον θα έπρεπε να κάνουμε μία έκκληση να προσθεθεί μία παράγραφος σχετικά με μικρότερα ε, ελάσσονο σημασίας αξιόπινες πράξεις οι οποίες δεν πρέπει να περιληφθούν σε αυτό το έγγραφο διότι υπάρχει πάντοτε το πρόβλημα και είναι ένα γενικό πρόβλημα το οποίο αναφέρουμε συχνά ότι υπάρχει το πρόβλημα της αμοιβαία αναγνώρισης και των αναγνωρισμένων ελαχίστων προδιαγραφών οπότε ε, πρέπει να υπάρχει ένας πολύ στενά περιγεγραμμένος πυρήνας ε, και ιδίως οι λόγοι για την ε, ε, απέλαση θα πρέπει να αναφέρεται δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διότι δεν πρέπει να επιτρέπεται για επουσιώδη αδικήματα αλλά πρέπει να υπάρχει και η αρχή της αναλογικότητας που θα λάβουμε υπόψη. Επίσης σε θέματα ευαίσθητα σε ε, παραδείγματος χάρη περιπτώσεις τηλεφωνικής παρακολούθησης πρέπει να δούμε αν είναι κάτι που πρέπει να ρυθμιστεί εδώ ή αν δεν θα έπρεπε να εξαιρεθεί και να λυθεί από κοινού με άλλα προβλήματα διότι όπως σας είπα η βάση αυτού του νομοθετήματος πρέπει να είναι πολύ περιορισμένη και να μην προσπαθήσουμε όλα να τα ρυθμίσουμε συλλήβδιν εδώ. Όπου λοιπόν δεν υπάρχουν προβλήματα και όπου είναι σαφής η αρχή της αναλογικότητος, άπαξ και επιθυμούμε να θεσπίσουμε αυτό το μέτρο, θα πρέπει να προχωρήσουμε και μετά να δούμε εάν μπορούμε να στραφούμε στα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο για να καταρτιστούν ελάχιστες προδιαγραφές. Οπότε ο καθένας θα μπορέσει να ε, καταλάβει ότι το κοινοβούλιο Βούλιο δίνει ένα σαφνό, σαφές μέτρο ότι θέλει αυτή την ρύθμιση αλλά θέλει συγχρόνως να καταρτιστούν ελάχιστες προϋποθέσεις πράγμα που έχει γίνει προς το παρόν για τους δικηγόρους και για τους εισαγγελείς και από πλευράς δικηγόρων. Νομίζω ότι η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών είναι σημαντική και πρέπει να ισχύσουν οι, τα ίδια δικαιώματα και οι ίδιες δυνατότητες για την <clears throat> υπεράσπιση και να υπάρχει μια ισορροπία. Λοιπόν, ελπίζω ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε μια κοινή απόφαση. Ευχαριστώ. <clears throat> Ο κύριο Μπρόνς. Δεν ξέρω αν κάτι δεν κατάλαβα καλά, αλλά σήμερα το απόγευμα είχα καταλάβει ότι ακούσαμε πως εάν ε, το αδίκημα της πρώτης χώρας δεν ήταν αδίκημα στη δεύτερη χώρα, τότε η δεύτερη χώρα μπορεί να έχει το δικαίωμα να μην αναγνωρίσει το αίτημα και άρα να μην εκτελέσει την έρευνα. Αυτό όμως αντιβαίνει στους κανόνες του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, όπου ένα ένταλμα ε, σύλληψης ε, ισχύει και στη δεύτερη χώρα, παρόλο που το δίκημα μπορεί να μην θεωρείται δίκημα στη δεύτερη χώρα. Δεν υπάρχει αντίφαση λοιπόν, γιατί οι αρχές της πρώτης χώρας μπορούν να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης επειδή υπάρχει υποψία για αδίκημα στην πρώτη χώρα που δεν είναι αδίκημα στη δεύτερη χώρα. Η δεύτερη χώρα όμως πρέπει να εκτελέσει, δεν ξέρω αν ε, σας έκανα να μπερδευτείτε. Εγώ πάντως είμαι κατά της ε, έκδοσης από μια χώρα στην οποία δεν είναι αδίκημα εκείνο για το οποίο έχει ζητηθεί η έρευνα. Πάντως έτσι κι υπάρχει εδώ πέρα αντίφαση. Γιατί τελικά καταλήγουμε στο τι, ζητάμε η δεύτερη χώρα να εκδώσει κάποιον για ένα δίκημα το οποίο δεν είναι δίκημα σε εκείνη τη χώρα, τη δεύτερη. Ο κύριος Κοέλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω τις ε, ανησυχίες που εξέφρασε ο εισηγητής Νούνο Μέλο όσον αφορά την Ευρώπη ως χώρο δικαιοσύνης. Πολλοί από εμά εδώ, σε αυτή την αίθουσα και στην Ολομέλεια, είπαμε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μόνο η Ευρώπη της ασφάλειας, αλλά να είναι και η Ευρώπη της δικαιοσύνης. Και θέλουμε αυτό να το προωθήσουμε με την, ε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας, αλλά και με κάποια μικρά βήματα ε, Ωστόσο πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν για να ενισχυθεί αυτό που έλεγε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, δηλαδή είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη, ο ακρογωνιαίος λήθος δηλαδή της ε, συνεργασίας. Πιστεύω πως η έκθεση του Νούνο Μέλο ανταποκρίνεται σε κάποιες από τις ανησυχίες και θα μπορούσαμε να έχουμε σε σχέση με την ενίσχυση της συνεργασίας ε, και στην έρευνα στα ποινικά αδικήματα. Αυτό που θέλουμε οπωσδήποτε, ε, μάλλον το πολύ σημαντικό θέμα είναι η νομιμότητα και σχετίζεται με την προστασία των δικαιωμάτων και αυτό είναι κάτι που ε, αναφέρεται σωστά στην έκθεση του κυρίου Μέλου. Εκτιμώ τις αναφορές στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και όπως είπε και ο συνάδελφος ε, Κροτσέτα, είναι υποχρεωτική η παρέμβαση μιας δικαστικής αρχής. Είναι αυτό πολύ κρίσιμο ακριβώς για να αυξηθεί η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, πως ξεκινάμε σωστά αυτή τη διαδικασία στο πλαίσιο της συναπόφασης που θα μας υποχρεώσει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια συνεργασίας ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο. Ο κύριος Φως. Χαίρομαι λόγω του φιλόδοξου σχεδίου εκθέσεως και συγχαίρω τον εισηγητή για ε, την προσπάθεια εναρμονίσεως της ε, ποινική συνεργασίας και ε, πριν από την προετοιμασία δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω το κείμενο αλλά μπορώ τώρα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες έχω σημειώσει και τις οποίες έχω ήδη αναφέρει. Καταρχήν βρίσκω ότι οι διάφορες νομικές διατάξεις και οι ε, οι παραδόσεις μεταξύ κρατών μελών είναι πάρα πολύ σωστές και χαίρομαι για την αρχή της ε, αναλογικότητος ε, και για τη μνήα της ε, τόσο στο προήμιο όσο και στο άρθρο 5α διότι υπάρχουν πολλά κράτη που έχουν ανάγκη κάτι τέτοιο και στο κράτος εκτελέσεως βεβαίως δέχεται να υπάρξει μία παραβίαση αυτής της αρχής πράγμα που δεν επιτρέπεται και παραπέμπουμε στην παράγραφο 9 στο καινούριο άρθρο 5α. Χαίρομαι και για την επιφύλαξη του δικαστή, πράγμα το οποίο θεωρώ απαραίτητο και στο άρθρο 17 θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό το, το, κείμενο που διατυπώθηκε και, και όσον αφορά το ο Πέλλας είναι λέγγι ε, θεωρώ ότι και αυτό είναι χρήσιμο χωρίς να είμαι βέβαιος ο, αν καλύπτει όλες τις ανάγκες και το 3-7 ή στο άρθρο 10 το 3 και το 7 θα έπρεπε ίσως να επανεξεταστούν. Ε, πέραν αυτού κάθε άλλος λόγος της παραπομπής μπορεί να θεωρηθεί ότι ε, αναστρέφει την ισορροπία και θα πρέπει να κοιτάξουμε ε, στις σχέσεις μεταξύ των κρατών ε, να μην αναφερόμαστε σε τάξεις οι οποίες είναι πεπερασμένες και να κοιτάξουμε να προχωρήσουμε. Όσον αφορά την την ημερομηνία καταθέσεως των τροπολογιών είναι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, μακρύτερος χώρος, χρόνος από ό,τι συνήθως, αλλά πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα με πολύ ευαίσθητο περιεχόμενο και γι' αυτό θα έπρεπε να κοιτάξουμε να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο ώστε να έχουμε άλλη μία ανταλλαγή απόψεων κατά τρόπον ώστε να το εξετάσουμε λεπτομερώς, να το ξαναδιαβάσουμε με προσοχή και γι' αυτό θα ζητούσα η προθεσμία να μετατεθεί ακόμη μακρύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Ιντβελτ. Ευχαριστώ. Η Σκιώδη, η Βαρονιλάτ Λάτφορτ, μου ζήτησε να μοιραστώ κάποιε ιδέε τη μαζί σα. Θα τα διαβάσω όμως. Λέει ότι χαίρεται για την πρόταση επί της αρχής. Λέει όμως ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν λάβουμε υπόψη μας τις εμπειρίες που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από αυτά που είχαμε προβλέψει. Επίσης υπογραμμίζει ότι πρέπει να περιλαμβάνονται τα δικαιώματα των υπόπτων βασιζόμενοι στην διαδικασία που ισχύει αλλά αναφέρεται επίσης και στη νέα προτινόμενη οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων. Για το θέμα της άρνησης ε, πρέπει να παραμείνει αρκετά ευρύ το θέμα αυτό και ότι πρέπει την άρνηση και την κάλυψη της έρευνας να είναι πράγματα τα οποία θα εξετάζουμε πολύ πριν αποφασίσουμε. Επίσης λέει ότι το θέμα της έκδοσης ε, αίτησης έρευνας λέει η κυρία Λάτφορντ ότι η πρόταση ε, του συγητή στην παράγραφο 22 για την εκτελεστική αρχή ότι πρέπει ε, το ότι λέει δηλαδή ότι πρέπει να είναι δικαστική αρχή θεωρεί η κυρία Λάτφορντ ότι δεν είναι αναγκαίο αυτό. Δικαστικές αρχές πρέπει να έχουν την ευθύνη του αιτήματο, ε, δηλαδή της έκδοσης του αιτήματο. Επίσης, όσον αφορά ε, τα επιχειρήματα για την άρνηση, να μην υπάρχει δυτή εγκληματικότητα ή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εδώ η κυρία Λάτφορντ έχει κάποιες προτάσεις για την διατύπωση. Τέλος, Το άρθρο 13 έχει βελτιωθεί γιατί όντω έχουμε εμπνευστεί από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Θα έπρεπε όμω να δούμε μήπω το άρθρο αυτό μπορεί να γίνει πιο αυστηρό ακόμα, ιδιαίτερα για τους δικηγόρους να μπορούν να ζητούν τη μεταφορά αποδεικτικών στοιχείων βάσει της εντολής αυτής της ευρωπαϊκής έρευνας. Αυτά νομίζω. Εντάξει, έχει κι άλλα, αλλά καλύτερα διμερώς να τα συζητήσει με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλος το λόγο για το σημείο αυτό στην εμερήσια διάταξη, οπότε το λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Μέλο. Ο κύριος Κορτσέτο κάτι έχει να πει, να προσθέσει. Συμφωνώ με την πρόταση για την αναβολή της ε, ημερομηνίας υποβολής των ε, τροπολογιών. Πιστεύω ότι 31 ήταν πολύ κοντά. Μήπως μπορούσαμε να πάμε τουλάχιστον μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου, γιατί 31 πέφτει η Τρίτη. 3 Φεβρουαρίου είναι η Παρασκευή, δηλαδή στην ουσία κερδίζουμε μια εβδομάδα δουλειάς. Φαίνεται να είναι μόνο τρεις μέρες, αλλά στην ουσία είναι μια εβδομάδα εργασίας που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Ευχαριστούμε κύριε Κροτζέτα. Πριν δώσω πάλι το λόγο στον κύριο Μέλο, η γραμματεία μου είπε πω είναι δυνατόν να παρατείνουμε την, υπο... την προθεσμία υποβολή τροπολογιών και θα σα την ανακοινώσουμε εάν συμφωνείτε κι εσεί. Οπότε τώρα δίνω το λόγο σε εσά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να πω ότι κατέγραψα με μεγάλη χαρά την ε, βασική συνένεση που είδαμε να επικρατεί με βάση όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν και πάλι και τη συμφωνία του Συμβουλίου και της ε, Κομισιόν. Παραμένουν κάποιες ανησυχίες του κύριου Κροτσέτα Βεβαίω, ε, πριν από λίγο καιρό διανεμήθηκε η έκθεση, αλλά νομίζω πω αυτέ οι ανησυχίε σα καλύπτονται στι τροπολογίε που έχουν υποβληθεί. Για παράδειγμα, όταν είπατε ότι το ένταλμα θα πρέπει να εκδίδεται από κάποιον εισαγγελέα. Προβλέπετε, Μόλι αυτό κάναμε, να, είναι, να μην είναι δηλαδή κάποια αστυνομική αρχή που θα καθορίζει ότι ο εισαγγελέα κάποια άλλες χώρα θα πρέπει να εκδώσει ε, ένταλμα. Όχι, θα πρέπει να γίνεται από του εισαγγελεί των ε, ενδιαφερόμενων χωρών. Επίσης, ε, αυτό που είπατε, ότι ποιος ε, επικυρώνει την εγκληματική, τον εγκληματικό χαρακτήρα μιας πράξης ή όχι. Θα πρέπει να είναι η χώρα εκδοσής αλλά και η χώρα παραλαβής αν δεν θεωρείται αδίκημο θα πρέπει να υπάρχει αίτημα ε, και μπορεί ωστόσο η χώρα που το λαμβάνει να μην προβεί στην παράδοση των αποδείξεων αν τα στοιχεία δεν δίνουν ε, ε, δεν στοιχειοθετούν αδίκημα για την ίδια τη χώρα αυτή. Και για την υπεράσπιση είναι πολύ σημαντικό, όντως εγώ είμαι δικηγόρος ο ίδιος. Υπάρχει το βασικό δικαίωμα υπεράσπισης σε οποιαδήποτε χώρα δικαίου που θέλει να ονομα, αποκαλείται κράτος δικαίου. θα πρέπει να γίνεται κάποια παρέμβαση σε, στην έδρα της προσφυγής, εκεί όπου γίνεται δηλαδή η καταγγελία και Επίσης, συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Ιντεφέλντα όσον αφορά τη δυνατότητα των, ε, των ε, νομικών να ζητήσουν ε, ένταλμα ή δράση. Προβλέπεται στο άρθρο 13, προβλέπεται αυτό, όταν λέει ότι οι αρχές της χώρας έκδοσης και της χώρας παραλαβής των, των μπλεκόμενων χωρών, της μιας και της άλλης δηλαδή, αυτές δίνουν στους ενδιαφερομένους τις κατάλληλες ε, ε, πληροφορίες ώστε να εγγυηθούν την ουσιαστική άσκηση του ε, δικαίου, όπως προβλέπεται η πραγματική άσκηση του δικαιώματο προσφυγή και του δικαιώματο δράση που προβλέπονται στι προηγούμενε παραγράφου. Σημαίνει δηλαδή ότι μπορούν ε, να χρησιμοποιηθούν για, με μεγαλύτερο εύρο όπω αυτό συμβαίνει σε, κάποιο, σε οποιαδήποτε κράτο δικαίου. Και σε σχέση με τις παρατηρήσεις του κυρίου Άλμπρεχτ, τον ευχαριστώ επίση για τα σχόλιά του, να, να του πω ότι Το παράδειγμα που αναφέρατε ήδη αποτελεί συγκεκριμένο λόγο κατηγορίας. Ας πούμε, ένας δικαστής Πορτογάλος ζητά έρευνα στην Γερμανία, αλλά τα στοιχεία που αιτιολογούν ε, αυτό το αίτημα δεν ε, στοιχειοθετούν αδίκημα στη Γερμανία, μπορεί η Γερμανία να αρνηθεί το αίτημα. Αυτό προβλέπεται. Ο κύριος Μπρόντς με ρώτησε σε σχέση με το θεσμό της έκδοσης σε αντίθεση με την ε, ποινική έρευνα. Δεν ξέρω αν δεν σας κατάλαβα καλά. Ελπίζω να μην σας παρανόησα. Μια χώρα μπορεί να μην προβεί στη δράση σε σχέση με την παροχή των αποδείξεων αν τα στοιχεία, <coughs> αν τα στοιχεία δεν στοιχειοθετούν αδίκημα στη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό ε, δεν έρχεται σε αντίθεση με τον θεσμό της έκδοσης γιατί μπορεί μια χώρα να αρνηθεί την έκδοση και επί τη βάση της εθνικής τους ε, ε, νομοθεσίας αλλά και επί τη βάση κάποιων ετοιμάτων. Ας πούμε η Πορτογαλία δεν εκδίδει έναν πολίτη αν το αδίκημα είναι ένα αδίκημα το οποίο επισύρει θανατική ποινή σε άλλη χώρα, στην άλλη χώρα. Μπορεί να στοιχειοθετούν έγκλημα στην τάδε, στη ΣΥΠΑ, π.χ. Εντάξει, εδώ είμαστε, δεν είμαστε σε αυτό το πλαίσιο γιατί είναι χώρα εκτός της Ένωσης. Αλλά ας πούμε για μια χώρα όπου ισχύει η θανατική ποινή, αν τη ζητηθεί της Πορτογαλίας να εκδώσει κάποιον πολίτη, δεν πρόκειται να τον εκδώσει. Αυτό σας το λέω για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο ένταλμα έρευνας και την έκδοση. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εδώ, μιλάμε, εδώ λέμε ότι το ένταλμα έρευνα μπορεί μια χώρα να το αρνηθεί, να το απορρίψει, από τη στιγμή που τα στοιχεία που τις διαθέτει ο εισαγγελής, ο εισαγγελέας δεν στοιχειοθετούν ε, αδίκημα. Μπορούμε να το συζητήσουμε και μεταξύ μας για να το συνονοηθούμε καλύτερα. Ε, Όσον αφορά τις προθεσμίες δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όλοι μας κερδίζουμε νομίζω να έχουμε μια πιο μεγάλη προθεσμία ώστε όλοι να μπορέσουμε να μελετήσουμε τα συντάγματα και το, σε νομικές προβλέψεις, ούτως ή άλλως θα ξαναειδωθούμε στα Στρασβούργο με τους σκιώδεις εισηγητές και μπορούμε να το εξετάσουμε μαζί εκεί το θέμα, αλλά ούτως ή άλλως δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραταθεί η προθεσμία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μέλο. Και τώρα έρχομαι στο δεύτερο σημείο της σημερινής διάταξης για απόψε που αναφέρεται στην κατάσταση στην Ουγγαρία. Έχουμε εδώ μεταξύ μας την κυρία Φρανσουάζ Λεμπάλ, να της δώσω δύο λεπτά να έρθει εδώ στο έδρανο της Προεδρίας. Είναι Γενική Διευθύντρια για τη, της Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και θα μας παρουσιάσει την έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Αυτό το θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη μετά από αίτημα των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων. Uh, Θα δώσουμε το λόγο τώρα, πρώτα στην κυρία Ντεμπάιλ και μετά σε όσους ευρωβουλευτές, συντονιστές και λοιπά που θέλουν να μιλήσουν εκ μέρους των πολιτικών ομάδων και μετά στους υπόλοιπους. Τι θέλετε? Κύριε Πρόεδρε, είμαι Ουγγαρέζα στους μη αγεγραμμένους. Είμαι και δικηγόρος και θέλω να είμαι βεβαίω ότι θα πάρω το λόγο κάποια στιγμή. Ναι, ναι, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα εσείς κύριε Αντεμπάλη ενημερώστε μας για την κατάσταση πώς έχει, τη λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας εδώ. Και αυτό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδρασε αμέσως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλιστα και πριν από οποιοδήποτε άλλον και εξέφρασε την θέση της πολύ γρήγορα πριν δημοσιευθεί η σχετική νομοθεσία, πριν αρχίσει να ισχύει δηλαδή το νέο σύνταγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μία νομική άποψη βέβαια. Είναι θεματοφύλακας των ε, συνθήκων η Κομισιόν και βάσει αυτού λοιπόν η Κομισιόν αξιολογεί το κατά πόσο συμμορφώνεται η Ουγγρική νομοθεσία με την κοινοτική νομοθεσία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εκφράστηκε ήδη από την Επίτροπο Ρέντινγκ από το Δεκέμβριο με επιστολή της προς τον κύριο και Υπουργό Δικαιοσύνης, όπου εκφράστηκαν οι κύριες ανησυχίες μας. Πρώτον, στο θέμα της δικαιοσύνης, γιατί εδώ μιλάω για την δικαιοσύνη βασικά. Λοιπόν, μία από τις κύριες ανησυχίες εδώ είναι η ηλικία συνταξιδότηση των δικαστών και των εισαγγελέων. Με το νέο Ουγγρικό Σύνταγμα με εξαίρεση του Προέδρου του Κούρια κανένας δικαστής ή εισαγγελέα δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 62 που είναι ηλικία συνταξιοδότησης. Έτσι, από τα 70 που ήταν τώρα ηλικία συνταξιοδότησης των δικαστών κατεβαίνει στα 62. Και Έτσι λοιπόν, θα 31 Δεκεμβρίου πρέπει να συνταξιοδοτηθούν όσοι δικαστές είναι πάνω από το όριο αυτό. Τι κοιτάζει και τι εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε αυτό. Κατά πόσο είναι συμβατό το μέτρο αυτό με την οδηγία ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την απασχόληση. Η οδηγία αυτή και είναι 274 δικαστές αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αποχωρήσουν. Έτσι λοιπόν, αν φανεί ότι υπάρχει διάκριση, η διάκριση αυτή θα πρέπει να γίνεται με κάποια αντικειμενική και αναλογική αιτιολόγηση. Στην περίπτωση του ογκρικού νόμου η κατάσταση είναι και πιο σοβαρή νομικά ακόμα επειδή η κυβέρνηση δήλωσε ότι θέλει την ηλικία συνταξιοδότησης να την πάει από 62 στα 65 τις επόμενες χρονιές. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο και δεν ακούγεται, ακούγονται παράσιτα. Ας μικρόφωνο. Όχι, ακούγονται πολλά παράσιτα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε.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 Okay. Uh, is it better? Then I would be glad to offer it to... Δοκιμάζουν όλα τα μικρόφωνα, αλλά όχι, δυστυχώς υπάρχει το ίδιο πρόβλημα με όλα τα μικρόφωνα από το Προεδρείο.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 Now, I'm sorry. Now, please continue. Yes, Φαίνεται ότι διορθώθηκε. Ναι, διορθώθηκε το πρόβλημα. Πού ήμουνα λοιπόν. Και για να βγαίνει καλά στην εικόνα πρέπει να χρησιμοποιεί το αριστερό μικρόφωνο η ομιλήτρια. Γι' αυτό και αλλάζει. Ωραία. Τι έλεγα λοιπόν. Έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να δει κατά πόσο η νομοθεσία της Ουγγαρίας ευθυγραμμίζεται με τις κοινοτικές προδιαγραφές και σε θέματα που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη υπάρχουν τρία σημεία ανησυχία. Το πρώτο σημείο ανησυχία, όπως εξηγούσα, είναι η ηλικία σταξιοδότηση των δικαστών και εισαγγελέων. Πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι συμβατά τα μέτρα αυτά, τα οποία μειώνουν τη ταξιδότηση των δικαστών από τα 70 στα 62, να δούμε κατά πόσο αυτό το μέτρο είναι συμβατό με την οδηγία για την ίση μεταχείριση και απασχόληση και να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει διάκριση σε βάρος αυτών των ε, ατόμων. Μάλιστα την ίδια στιγμή που η ίδια εγκρική κυβέρνηση σκέφτεται να αυξήσει το όριο ταξιοδότησης από τα 62 στα 65. Και όπως ε, έλεγα, 274 δικαστές θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν στις 31 Δεκεμβρίου του 2012. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος τομέας ανησυχίας μας. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Σύμφωνα με την νομοθεσία, η Προεδρία του νέου ε, Εθνικού Δικαστικού, της Νέας Δικαστικής Υπηρεσίας όσον αφορά την ε, λειτουργία των δικαστηρίων, όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, τον προπολογισμό κτλ. Είναι αρμόδιο αυτός, ο επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής. Δηλαδή εκείνος από μόνος του παίρνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις για το δικαστικό σώμα. Δεν υπάρχει δηλαδή συλλογική απόφαση όσον αφορά τη λειτουργία των δικαστηρίων. Επιπλέον, η εντολή του τέος Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου εξελέγει για έξι χρόνια, το 2009, και ολοκληρώνεται το 2011, σε αντίθεση με άλλους δικαστές από το Ανώτατο Αυτό Δικαστήριο, εκείνοι συνεχίζουν την εντολή τους ως δικαστές του νέου Κούρια, που αντικαθιστά το Ανώτατο Δικαστήριο. Τέτοια συγκέντρωση εξουσιών και η πρόορη πάυση της εντολής του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου θέτουν το ζήτημα της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος. Και το κατά πόσο είναι συμβατά τα μέτρα αυτά με το άρθρο 47 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι ένα θέμα που εξετάζουμε. Το εξετάζουμε μια από το άρθρο 47 λέει ότι Όποιανού τα δικαιώματα διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παραβιάζονται, έχει το δικαίωμα διόρθωσης από έναν εξάρτητο δικαστήριο. Και αυτό έχει να κάνει με οποιαδήποτε κατηγορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, τίθονται συστηματικά ζητήματα που πρέπει να ελέγξουμε όσον αφορά αυτή την νομοθεσία. Πάντα για τον ε, τομέα τώρα το δικαστικό. Το τρίτο στοιχείο ανησυχίας που εκφράζει και η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ στον Υπουργό Ναβράτσικ έχει να κάνει με την ανεξαρτησία της του επόπτη προστασίας δεδομένων. Σύμφωνα με την ένομο νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, η Εθνική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων, που αντικαθιστά αντικαθιστά την υπηρεσία της Επιτροπής για την Προστασία Δεδομένων. Η νομοθεσία αυτή λοιπόν έπαυσε πρόωρα την εντολή, την εξάχρονη κανονικά, του Επιτρόπου για, τα, για την προστασία δεδομένων, ο οποίος είχε οριστεί το 2008. Επιπλέον η νομοθεσία αυτή προβλέπει την δυνατότητα απόφασης απόλυσης από τον Πρωθυπουργό ή από τον Πρόεδρο. Βάσει αυθαίρετης απαλλαγής. Το συμβατό ή όχι του μέτρου αυτού με την αρχή της ανεξαρτησίας των Εθνικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων που ισχύει από το 1996 και με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι βέβαια κάτι που επίσης μας απασχολεί. Επιπλέον από τις ανησυχίες αυτές στον τομέα της δικαιοσύνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες και για κάποια άλλα θέματα, ιδιαίτερα για το θέμα της ανεξαρτησίας της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Ουγγαρίας δηλαδή, κάτι σχετικά με το οποίο εκφράστηκε η Αντιπρόεδρος νωρίτερα. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι σημαντικό τώρα είναι να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τη νομική της ανάλυση, γιατί ως θεματοφύλακας των συνθήκων πρέπει να βασίζεται σε νομικά στοιχεία. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα ολοκληρώσουν την ανάλυση τους έγκαιρα ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να αποφασίσει την επόμενη εβδομάδα στην συνάντησή της στις 17 δηλαδή Ιανουαρίου. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει πλήρως τα προνόμια της ως θεματοφύλακα των συνθήκων και ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που έχει προσφυγής επί στην περίπτωση που έχει αρκετές νομικές αποδείξεις ώστε να μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Και ελπίζουμε ότι η Ουγγαρία θα το δεχτεί ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή λοιπόν θα αποφασίσει τι ακριβώς δράση θα αναλάβει αφού ολοκληρώσει την ανάλυση της αυτή την επόμενη εβδομάδα στις 17 του μηνός θα πάρει την απόφασή της η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Κυρία Λεμπέλ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε. Στρέφομαι τώρα προς τους συναδέρφους, να δούμε ποιος θέλει το λόγο. Έχουν γραφτεί πολύ ήδη. Οπότε, πρώτα θα δώσω το λόγο σε όσους μιλήσουν εκ μέρους των ομάδων τους, που είναι δηλαδή συντονιστές οι ίδιοι, και μετά θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ να περιοριστείτε σε τρία λεπτά, όχι παραπάνω, γιατί τελείως δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Πρώτος, εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Έγγελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω να αφιερώσω την πρώτη μου παρθενική παρέμβαση σε αυτήν την Επιτροπή ε, σε κάτι πιο νομικό, κάτι πιο ουσιαστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού αυτή είναι η συζήτηση θα μιλήσω για αυτό το θέμα. Δεν θέλω να επεκταθώ στα όσα είπε ήδη η κυρία Λεμπάγε. Ίσως θα είχε νόημα να ασχοληθούμε με αυτό που διαδικαστικά γίνεται και με το ποιο μπορεί να είναι το πολιτικό υπόβαθρο των όσων συμβαίνουν. Από τότε που έγιναν οι ογκρικές εκλογές το 2010 κυβερνάτε ένα, ε, η Ουγγαρία από ένα κόμμα που πήρε το 53% ε, των ψήφων που του δίνει τα 2 τρίτα των εδρών στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο που είναι η πλειοψηφία που χρειάζεται για να προχωρήσει μόνο του το κόμμα αυτό σε αλλαγές ε, του συντάγματος. Αυτό είναι ένα γεγονός, δεν αμφισβητείται αυτό από οποιονδήποτε και Ίσως να ακούγεται παράξενο που από καιρού εις καιρό έχει κανείς την εντύπωση πως ακόμα και αυτό θα πρέπει να αμφισβητηθεί, ότι είναι δηλαδή κάτι το παράνομο. Αυτή ήταν η βούληση των Ούγγρων ε, ε, ψηφοφόρων ε, το 2010. Η πλειοψηφία λοιπόν αυτή προχώρησε στην αλλαγή του συντάγματος, στη ριζική αλλαγή του συντάγματος. Ε, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο αλλού. Επίσης, επειδή ήταν δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, πόσο θυμάμαι, αυτό το σύνταγμα, ακόμα κι αν δεν ήταν ε, ομόφωνα αποδεκτό από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, εν γέννη συνοδεύθηκε από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, ψηφίστηκε από μια μεγάλη πλειοψηφία Ούγγρων ε, ε, ψηφοφόρων, 11% εξ αυτών, εξ αυτών εξέφρασαν την σύμφωνη τους νόμη και τώρα έχει μπει σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου το Σύνταγμα αυτό. Σύνταγμα λοιπόν και βασικές νομοθεσίες και τα προβλήματα που έθιξε η κυρία Λεμπάη, δηλαδή ε, ηλικία συνταξιδότηση των ε, δικαστών, ανεξαρτησία του δικαστικού σώματο, εκλογικό νόμο θα μπορούσα να προσθέσω εγώ που είναι υπό εξέταση αυτή τη στιγμή. Ε, νόμος περιθρησκειός και ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας που δεν εμπίπτει στην εντολή αυτής της Επιτροπής και γι' αυτό το λόγο μάλλον δεν το προσεγγίζουμε. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το θίξουμε σε διαφορετικό πλαίσιο. Από όσο γνωρίζω λοιπόν, είμαστε τώρα σε μια διαδικασία που προβλέπουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε περίπτωση που προκύψουν αμφιβολίες σε σχέση με τη συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ερευνά, όπως είναι καθήκον της και αρμοδιότητά της ως θεματοφύλακα των συνθηκών. Κατά πόσο δηλαδή τα νομικά μέσα που ψηφίζονται σε κάποιο ε, κοινοβούλιο κράτους μέλους είναι συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία ή όχι. Και θα έχουμε αυτή την αξιολόγηση της Κομισιόν την επόμενη εβδομάδα. Η Επίτροπος Ρέντινγκ ε, τη μίλησα μαζί της στο τηλέφωνο για να της ρωτήσω κάποιες πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Δεν έχω την εντύπωση πως η Επίτροπη δεν ξέρει τι κάνει. Αντιθέτως, ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Και Έχουμε δέσμευση από πλευρά των Ουγγρικών αρχών που έχει επαναληφθεί τις τελευταίες μέρες όχι μόνο για σοβαρή εξέταση των όσων θα συστήσει η Επιτροπή, αλλά και για το ότι θα ενεργήσει αντίστοιχα, όπως ήδη έχει κάνει εξάλλου, σε σχέση με το νομοθεσία περί ελευθεροτυπίας που επίσης προσέλκυσε την προσοχή του Κοινοβουλίου. Είναι εντύπωσή μου λοιπόν και εντύπωση του ΕΛΚ πως αυτή τη στιγμή θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική αξιολόγηση της Επιτροπής για το θέμα του Ουγγρικής νομοθεσίας. Θα έχουμε τα αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα και μετά θα δούμε τι θα προτείνει η Κομισιόν στις Ουγγρικές Αρχές και πώς αυτές θα αντιδράσουν. Από ό,τι φαίνεται οι Ουγγρικές Αρχές θα δεχτούν τα όσα θα τους προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ευθυγραμμιστεί αν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Και άρα θα ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά Εν τω μεταξύ δεν νομίζω ότι πρέπει να επικρατήσει ιστερία και δεν βλέπω γιατί εμείς εδώ, αυτή την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λειτουργήσουμε ως τελευταίο δικαστήριο, ως ε, ε, εφετείο κατά κάποιο τρόπο. Οι Ουγγρικές Αρχές έχουν απαντήσει στα ερωτήματα της κυρίας Ρέντινγκ ήδη σε ένα έγγραφο που περιλαμβάνει, αποτελείται από 90 σελίδες. Από αυτό ε, συνάγω ότι είναι σοβαρή για όλα αυτά και οπότε, εφόσον και η Κομισιόν είναι σοβαρή, ε, ας ολοκληρωθεί η υπόθεση την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε κύριε Έγγελ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Γκέρεντς. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν θα πάω τόσο παλιά στο χρόνο, όπως ο κ. Έγκελ, θα ήθελα να επιμείνω για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας και είναι αλήθεια ότι τώρα η Επιτροπή ενήργησε ταχύτατα. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις ε, Περίμενα δηλαδή κάποια παραπάνω πράγματα από την έκθεσή σας. Ε, μία από αυτές ε, σχετίζεται με τις ε, δικές σας προσδοκίες για την Ουγγρική κυβέρνηση. Σε ανακοινωθέν τύπου εχθές λέγατε πολύ ωραία ότι το κράτος δικαίου, η ελευθεροτυπία, ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι οι καλύτερες εγγύσεις για την εμπιστοσύνη των πολιτών και για την εμπιστοσύνη των εταίρων. Άρα λοιπόν ο καλύτερος τρόπος για να αρθούν οι ανησυχίες θα ήταν η δράση από τις Ουγγρικές αρχές. Τι είδου ε, δράση θα αναμένατε από τις Ουγγρικές αρχές στην επόμενη εβδομάδα, γνωρίζοντας ότι την επόμενη εβδομάδα οι Επίτροποι θα λάβουν την απόφαση για το κατά πόσο θα προχωρήσουν ή όχι σε διαδικασία επιπαραβάση. Όλοι ελπίζουμε πως δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο, αλλά θα ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε ποιε είναι οι προσδοκίες σας. Άλλη μου ερώτηση ε, σχετίζεται με την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και την ανεξαρτησία του ε, Γραφείου Επόπτη των ε, Προστασίας των Δεδομένων. Εσείς ε, είπατε, μάλλον ρωτήσατε, πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι το τέλος της εντολής πριν το τέλος της κανονικής θητείας δεν αμφισβητεί την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος ή του επόπτη της αρχής μάλλον προστασίας των δεδομένων. Οι απαντήσεις που δίνονται από τον κύριο Ναύρατσετς σε αυτό το έγγραφο των 90 σελίδων Αυτές οι απαντήσεις ήταν ικανοποιητικές για την Επιτροπή. Θα ήταν πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν πραγματικά πιστεύετε πως αυτές οι απαντήσεις είναι αυτές που ε, χρειάζονταν. Η επόμενη ερώτησή μου επίσης σχετίζεται με αυτά. Δεν πιστεύετε ότι η επανάληψη τέτοιου είδους αναδιοργάνωσης των ε, ανεξαρτησίες αυτών των ανεξαρτήτων ε, θεσμών όπως ε, η αρχή προστασίας των δεδομένων και, του δικαστικού, και η αρχή του δικαστικού σώματος δεν νομίζετε πως είναι πιο συστημικά θέματα και που θα πρέπει να τα αναλύσετε κατά κάποιο τρόπο στο συγκεκριμένο πλαίσιο και ότι χρειάζονται περισσότερο πολιτικές απαντήσεις και όχι μόνο νομικές που κατά κάποιο τρόπο επιτίθεται στην ανεξάρτητο θεσμό της δημοκρατίας ή επιτίθεται στις ισορροπίες των δημοκρατικών θεσμών. Είναι μια πολύ παρόμοια διαδικασία που γίνεται. Επίσης θα ήθελα κάπως να κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν και να αναφερθώ στη συζήτηση περί της νομοθεσίας για τον τύπο πέρυσι. Ο κύριος Έγκελ ανέφερε ότι φαίνεται πως οι ουγγρικές αρχές φαίνεται να είναι πρόθυμες να αλλάξουν οτιδήποτε χρειαστεί. Αυτό που συνέβη όμως πέρυσι με το νομοθεσία περί ελευθεροτυπίας ήταν ε, κάποιες καλοπιστικές αλλαγές που δεν άλλαγαν την ουσία, άλλαζαν την ουσία της ε, νομοθεσίας, αυτό το είδος δηλαδή συγκέντρωσης ε, που ε, αποπειράθηκαν να επιτύχουν, ε, όπως και τώρα με την νομοθεσία περί του δικαστικού σώματος. Ξέρω, θα ήθελα να γνωρίζω αν η Κομισιόν ε, διερευνά ή αναλύει τις επιπτώσεις της νομοθεσίας περί τύπου γιατί αναφέρθηκε από την Επίτροπο Κρούς ότι όταν θα είναι πια η ορατή της εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας θα είναι πρόθυμη να αναλύσει τις επιπτώσεις, των αντίκτυπο της εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας. Και με τα χαρά θα ακούγαμε τέτοιου είδους ε, νέα την επόμενη εβδομάδα σε σχέση με την νομοθεσία αυτή περί ε, τύπου. Έπειτα, δόθηκε μια εναλλακτική απάντηση στην δική σας επιστολή από τρεις ε, ανεξάρτητους θεσμούς ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη δημοκρατία στην Ουγγαρία που απάντησαν στις ίδιες ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στην κυβέρνηση. Θα ήθελα να γνωρίζω αν λάβατε αυτές τις απαντήσεις, αν τις αναλύετε και αν τις λαμβάνετε υπόψη. Γιατί διαφέρουν από τις κυβερνητικές απαντήσεις, φυσικά. Επίσης να ρωτήσω αν αναλύεται τον εκλογικό νόμο και όλους τους σχετικούς νόμους με τις δίκαιες και ελεύθερες εκλογές, γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι νόμοι που σχετίζονται με όλα αυτά ή που χαλαρά συνδέονται με όλα αυτά, για να μην μιλήσουμε για την Εθνική Κεντρική Τράπεζα, που δεν είναι αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής. Τα υπόλοιπα θέματα είναι αρμοδιότητες πάνω κάτω αυτής της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βέμπερα. Ευχαριστώ <clears throat> κυρία Πρόεδρε, έχω ορισμένα σχόλια και μετά τρεις ή τέσσερις ερωτήσεις. <clears throat> Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, δεν διεκπεραιώνεται και διευθύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρία θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν τρία χωριστά σώματα, οπότε για την Επιτροπή δεν είναι θέμα επικοριτότητος. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν το, Κοινοβούλιο θεωρήσει κάποια δεδομένη στιγμή ότι πρέπει να κινηθεί, ε, το, η συνθήκη της Λισαβόνας του δίνει το δικαίωμα να το πράξει. Βέβαια ε, πάντοτε ε, είμαστε ε, ανοιχτοί στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά έχουμε και ορισμένες δυσάρεστες εκπλήξεις όπως ο νόμος για τα μέσα ενημέρωση στην Ουγγαρία, για τους Ρωμά στη Γαλλία όπου στο τέλος δεν μπορέσατε να ασχοληθείτε και να λύσετε το ουσιαστικό πρόβλημα, άρα υπάρχουν προβλήματα. Όσον αφορά η έκθεση, την έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να μην απευθυνθούν μόνο στα άρθρα που έχουν διαβάσει και στις, ε, ε, ε, στις επιστολές σχετικά με την έκθεση της Βενετίας αλλά να διαβάσουν την έκθεση της Βενετίας η οποία είναι πολύ διαφωτιστική για το τι γίνεται με το θέμα αυτό στην Ουγγαρία. Μπορώ να σας το στείλω άμα επιθυμείτε. Όσον αφορά τα ερωτήματα που θέσατε, ε, σε γενικές γραμμές, το ερώτημα ποια είναι η νομική βάση για να ξεκινήσει μία διαδικασία παραβίασης εάν δεν μας ικανοποιήσει οι απαντήσεις που θα δώσει η κυβέρνηση της Ουγγαρίας σχετικά με την ηλικία των δικαστών αναφέρεστε εις την οδηγία που απαγορεύει τις διακρίσεις να το δεχτούμε. Αλλά ξέρουμε ότι πάντοτε προβλέπεται μία μεταβατική περίοδο σε ένα σύνταγμα όταν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι γίνεται όμως με τα υπόλοιπα. Ποια είναι η νομική βράση για να ξεκινήσετε μία διαδικασία παραβίασης ε, αν ε, πάει στην Κούρια ή το ανώτατο δικαστήριο ή αυτά τα οποία αναφέρονται στο σημείο 2 και 3 γιατί από ό,τι ξέρω για να ξεκινήσει μία τέτοια διαδικασία χρειάζεστε ευρωπαϊκή νομοθεσία και είμαι περίεργη να δω ποια είναι αυτή. Και έτσι έρχομαι και στο επόμενο ερώτημά μου. Δηλαδή, δέστε την τεράστια διαφορά που και τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά τα οποία συζητάμε όταν μιλάμε για την πρόσβαση των χωρών και την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν συζητάμε για το τι γίνεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν υπάρχει λοιπόν νομοθεσία και η νομοθεσία αναφέρεται στα θέματα που θέσατε σχετικά με τα άλλα σημεία, δηλαδή την ηλικία και τον επόπτη για την προστασία των στοιχείων. Εξετάσετε το άρθρο 2, διότι αυτό ζήτησε από την αρχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε το άρθρο 2, που αναφέρεται στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί να υπάρχει ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά νομίζω ότι χίλιες φορές η κυρία Ρέντινγκ μας έχει πει ότι αυτό μπορεί μόνο να συνδυαστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Χρειάζομαι λοιπόν κάποια νομική εξήγηση από εσά και έχω και μία ακόμη ερώτηση και μετά θα σταματήσω. Τι θα γίνει σχετικά με τους βασικούς κανόνες που αναφέρεται επίσης και στο θέμα της εκθέσεως της ε, Βενετίας διότι αντιλαμβάνουμε ότι το σύστημα αυτό θα ισχύσει για πολλές εκατοντάδες ετών μέχρι δηλαδή κάτι να αλλάξει στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βέμπερ, ο κύριος Σταβάρες. Ευχαριστώ. Εγώ θα αρχίσω με, τα γενικά θέματα και έχω μόνο μία συγκεκριμένη ερώτηση διότι με κάλυψε η κυρία Βέμπερ η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο λειτουργούν βάσει διαφορετικών παραμέτρων και διαφορετικών νομιμοποιήσεων. Οπότε έχω να αναφερθώ σε διάφορα θέματα, αλλά γενικά νομίζω ότι την πρώτη φορά που συζητήσαμε ε, το θέμα του Ουγγρικού νόμου για τα μέσα ενημέρωσης, χαθήκαμε στις λεπτομέρειες, δηλαδή ε, σε τι μοιάζει η από τους νόμους περιτύπου των άλλων ε, κρατών μελών. Αλλά η συσσόρευση και ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων κατέστησαν την νομοθεσία αυτή πολύ επικίνδυνη. Αυτό γίνεται και εδώ. Μπορούμε να συζητήσουμε τους θεμελιώδεις νόμους, το, το σύνταγμα, τα, τις διατάξεις που προσθέτει περί του δικαστικού στόματος η Ουγγαρία, αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι τα στοιχεία οικονομικής, η ε, οικογενειακής ομοιότητος που παρουσιάζει αυτή η νομοθεσία. Δηλαδή διαγράφει γράφεται μία κίνηση, μία κατεύθυνση η οποία ανησυχεί το Κοινοβούλιο. Σε γενικές γραμμές λοιπόν πρέπει να πω ότι οι πολίτες είναι αυτοί που κάνουν αυτούς τους ελέγχους και το βλέπουμε στις αναφορές τις οποίες λαμβάνουμε στην Επιτροπή Αναφορών εδώ ότι ο λαός, οι άνθρωποι μας περιμένουν, μας ε, ε, ε, απαιτούν να ασχοληθούμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό συμπεριλαμβάνει και τους Ούγγρους πολίτες ε, και στο άρθρο 39 λέγεται ότι δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ ένα ε, κράτος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να επανέλθει στην κατάσταση η οποία υπήρχε πρώτης Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δηλαδή, ε, στη χώρα μου αυτό που έγινε πριν το 1974 θεωρώ ότι πρέπει να ισχύσει και για την Ουγγαρία και θα οπισθοχωρήσουν ε, αν ε, ισχύσει αυτή η νομοθεσία. Και απευθύνομαι εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως έκαναν και άλλοι συνάδελφοι. Θα ήθελε η κυρία Ντεράιτ να μας πει ποιο είναι το πνεύμα της προσχωρήσεως μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, μπορεί μία υποψήφια χώρα με τέτοια νομοθεσία να αντιμετωπίσει προβλήματα στην προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα ζητούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει για να μπορέσει να προσχωρήσει η χώρα. Και αν ναι, τότε το συμπέρασμα είναι σαφές. Τι θα κάνουμε με μια χώρα η οποία εντωμεταξύ ήδη είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι ευθύς. Και όπως είπε ο συνάδελφος από το ΕΛΚ, πάρα πολλοί Ουγγροί ψήφισαν το ΦΙΝΤΕΣ και ψήφισαν υπέρ ε, του συντάγματος. Αλλά η δημοκρατία σημαίνει όχι μόνο να κυβερνούν οι πλειοψηφίες, αλλά και να αλλάζουν και ενδέχεται βέβαια να το απεφάσισε αυτό μία πλειοψηφία και τι συνεπάγεται για τις επόμενες πλειοψηφίες δηλαδή να υπάρξει μία εξέλιξη η οποία υπήρξε σε άλλα κράτη αλλά μία χώρα παραδείγματο χάρη η οποία ανησυχεί για την βιωσιμότητα των οικονομιών μας δεν θα έπρεπε να ανησυχεί και για τη βιωσιμότητα των δημοκρατών διότι η δημοκρατία είναι επίσης ε, κάτι που πρέπει να επιτρέπει να υπάρχουν δημοκρατικές αλλαγές, διότι ακούω στους διαδρόμους να συζητιέται το άρθρο 7 που θεωρούν ότι είναι η ατομική βόμβα που θα χρησιμοποιήσουμε, ενδεχομένως, αλλά μιλάμε για το άρθρο 7 ε, παράγραφος 2. Η παράγραφος 1 όμως είναι μία διαδικασία που ξεκινά ένα πολιτικό διάλογο και μπορούμε να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να σχολιάσει τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα ενός κράτους και είναι κάτι το οποίο μας δίδεται η ευκαιρία να κάνουμε και που μας επιτρέπει η διαδικασία μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι πρόκειται να πράξουμε. Ευχαριστώ κύριε Ταβάρες. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης, τελευταίος ομιλητής εν ονόματι της πολιτικής ομάδος. Um, eh, Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ζητήσω όσοι δεν έχουν γραφτεί και αυτοί να μπορέσουν να πάρουν το λόγο στο πρώτο γύρο των εκπροσώπων των ομάδων. Είπατε πριν ότι τρία λεπτά έχει ο κάθε εκπρόσωπος της ε, ομάδας. Δεν έγινε όμως αυτό, κανένας δεν τήρησε το χρόνο του. Ο καθένας τους μίλησε πάνω από πέντε λεπτά. Και μετά βέβαια θα έχουμε λίγο χρόνο οι υπόλοιποι. Και στους άλλους θα δώσετε ένα ή μισό λεπτό. Θα ήθελα και αυτοί που δεν έχουν ε, γραφτεί για τον πρώτο γύρο και αυτοί έχουν τρία λεπτά στη διάθεσή τους. Όσοι δεν έχουν γραφτεί και αυτοί εκπροσωπούν κάποιους. Ευχαριστώ. Uh, Mr. Uh, we, uh, minutes. Τρία λεπτά είχα πει και όντως ήμουν αρκετά γενναιόδορη με τους συντονιστές και με τους εκπροσώπους των ομάδων. Μπορώ λοιπόν να πω ότι επειδή είστε από τους μη γεγραμμένους θα έχετε κι εσείς όντως τον ίδιο χρόνο πέντε λεπτά όπως ε, πήραν και οι προηγούμενοι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιος θα είναι εσείς. Α, ε, όχι εσείς. Όποιος όταν έρθει η σειρά σας Ξέρετε ότι στη Λίμπε συνήθω οι μη γεγραμμένοι δεν ε, παίρνουν το λόγο σε εκπρόσωποι ομάδων, αλλά συμφωνείτε τώρα με αυτή τη ρύθμιση. Ναι. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν, όπω είπαμε, από τι ομάδε ο κ. Στατεφλίδη. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάλυση που μας έκαναν ε, σήμερα. Νομίζω ότι είναι στο σωστό δρόμο και ότι η απόφαση που θα ληφθεί στις 17 έρχεται τη σωστή στιγμή. Από όσο ξέρω, πρόκειται να γίνει συζήτηση και στην Ολομέλεια εκείνη την ημέρα ή μια-δύο μέρες μετά. Συνεπώς θεωρώ ότι είναι πολύ καλό που θα ληφθεί απόφαση τότε. Τώρα, δεν γνωρίζω πόσα θέματα έχετε εξετάσει για να δείτε αν είναι συμβατά ή όχι με το κοινοτικό κεκτημένο. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, τα θέματα αυτά το θέμα της παραβίασης του εργασιακού δικαίου έχει εξεταστεί. Όχι μόνο δηλαδή το θέμα της ταξιοδότησης των δικαστών, αλλά γενικότερα κατά πόσο τα εργασιακά, οι εργασιακοί νόμοι τηρούνται ή όχι. Μήπως υπάρχει απειλή για τους οργανωμένους ε, εργαζόμενους. Ε, πράγματα γενικότερα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία. Ευχαριστώ. Θέλω και από αυτόν την άποψή σας. Ευχαριστούμε. Ερχόμαστε λοιπόν στο δεύτερο γύρο παρεμβάσεων. Τα απλά μέλη της Επιτροπής μας. Και θα σας δώσω το λόγο. Αλλά προηγουμένως, κύριε Σίπελ, κοιτάξτε συνάδελφοι, προσπαθήστε σας παρακαλώ δύο λεπτά ο καθένας προκειμένου να μπορέσουμε να τελειώσουμε έγκαιρα και να μπορέσουμε να ακούσουμε και την απάντηση της κυρίας Λεμπάιλ. Και όπως υποσχέθηκα βέβαια εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων θα έχετε εσείς πέντε λεπτά. Η κυρία Σίπολη λοιπόν πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που είπε στην αρχή η κυρία Λεμπάη, δηλαδή ότι η Επιτροπή είναι θεματοφύλαξ των συνθήκων και μετά πρόσθεσε ότι η Επιτροπή πρέπει να φροντίσει για να υπάρχει ακολούθηση και εφαρμογή των συνθήκων. Αλλά αυτό δεν επαρκεί γιατί στις διάφορες συνθήκες Μάστριχτ, Νικέας, Λισαβόνας έχουμε δεσμευτεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παραμένουν οι αρχές μας κοινέ, να υπάρχει ελευθερία, δημοκρατία, έλλειψη διακρίσεων και βλέπουμε ότι αυτά τώρα περιορίζονται και δεν ε, ελέγχονται επαρκώς με την εφαρμογή των νομοθεσίας. Πέρυσι λοιπόν η Επιτροπή καθυστέρησε για το θέμα του νομοθεσίας του τύπου γιατί στράφηκε ε, προς το Συμβούλιο και έπρεπε να έχει στραφεί και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως τότε δεν ήταν έτοιμο ε, διακομματικά να ε, κατά ε, να κατακρίνει τα μέτρα τα οποία έλαβε η Ουγγρική κυβέρνηση και υπάρχει ε, ένα θέμα σχέσεων μεταξύ Ουγγαρίας και, ε, και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν είμαστε ένα δικαστήριο αλλά εδώ συζητάμε παραδείγματος χάρη για την οικονομική κρίση και την κρίση του χρέους. Το θέμα είναι όμως ότι οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους και στους πολιτικούς χειρισμούς των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και έχουμε ε, πολλές ε, ε, νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες πότε είναι καλές πότε είναι ανεπαρκείς και πάντοτε μας απαντούν ότι είμαστε ε, μία κοινότητα έχουμε αλλαγές αλλά πρέπει να ισχύουν οι ίδιες αρχές και, τα, ε, και οι ίδιοι νόμοι και αυτό το καταρρύπτουμε με αυτά που γίνονται από την Ουγγρική κυβέρνηση και από το τι γίνεται ή δεν γίνεται ε, από τα ευρωπαϊκά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε πλέον να παραβλέψουμε ούτε να ωρεοποιήσουμε διότι και διεθνώς νομίζω ότι θα χάσουμε κάθε αξιοπιστία εάν σε όλα αυτά τα θέματα που ζητούμε από τους άλλους ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα εμείς τα ωρεοποιούμε και τα συγκαλύπτουμε στην Ευρώπη ε, διότι εάν θέλουμε να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Με συγχωρείτε πρέπει να σας σταματήσω τώρα, η κυρία Ιντφελτ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη γιατί λίγα έχω να προσθέσω στα όσα μόλις τόσο ωραία ακούσαμε από την κυρία Ζιμπελ. Θέλω όμως να απαντήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Έγκελς πρώτα απ' όλα, που είπε ότι η Ουγγαρία είναι κυρίαρχη χώρα και άρα μπορεί να αποφασίσει να κάνει ό,τι θέλει. Σας υπενθυμίζω ότι η Ουγγαρία, όπως και άλλες 26 χώρες, πήρε κυρίαρχα την απόφαση να υπογράψει την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάσει αυτής έχει κάποιες υποχρεώσεις. Αυτό που συζητάμε σήμερα δεν είναι η Ουγγαρία. Το πρόβλημα δεν είναι η Ουγγαρία. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη εφαρμογής του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών κανόνων του δημοκρατικού παιχνιδιού στην Ευρώπη. Και αυτό είναι τμήμα της ε, φάσης βάσει της οποίας οριμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση στην Ουγγαρία όντω είναι ιδιαίτερα σοβαρή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες μέλη που παραβιάζουν τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα Γι' αυτό και το σώμα μα έχει ζητήσει επανειλημμένω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει. Είτε πρόκειται για του Ρώμα στη Γαλλία που αναφέρθηκε, είτε πρόκειται για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, είτε πρόκειται για περιορισμό τη ελευθερία του τύπου, είτε πρόκειται για παραβιάσεις όσον αφορά του ζητούντε άσυλο όπω γίνεται στη δικιά μου τη χώρα. Ε, λοιπόν, έχουμε συμφωνίε συμβάσει και πρέπει αυτέ να εφαρμόζονται. Αυτό είναι το βασικό. Το ίδιο και στην Ευρωζώνη. Έχουμε ένα σύμφωνο σταθερότητα, το οποίο δεν είναι αξιόπιστο παρά μόνο αν τηρείται. Το ίδιο και για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ερώτηση λοιπόν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ απόλυτα με την Ρενάτε Βέμπερ για το ότι το σώμα μα είναι υπεύθυνο και έχει αυτόνομα το δικαίωμα να θέσει σε εφαρμογή ή όχι το άρθρο 7 και συγκεκριμένα το 7.1 της συνθήκης που δεν έχει να κάνει μόνο, δεν έχω βέβαια το κείμενο μπροστά μου, δεν έχει να κάνει μόνο με το κίνδυνο σοβαρής ε, παράβασης. Δηλαδή τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δίνουμε την ευκαιρία στο κράτος μέλος να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συζητήσει. Άρα δεν ε, εδώ πέρα διακόπτουμε τίποτα δικαιώματα. Τέλος. Μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερθήκατε σε τρεις τομείς ανησυχίας, όπως είπατε. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται και κάτι κάνει. Βέβαια, κατόπιν ερωτή, αφού άρχισαν να ισχύουν οι νόμοι αυτοί, υπάρχουν όμω και άλλοι τομεί ανησυχία. Ο νόμο για τα μέσα ενημέρωση. τι γίνεται εκεί. Ήδη έχει κλείσει ένα ραδιοφωνικό σταθμό, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι άλλο θέλει για να αρχίσει και εκεί να κάνει κάτι. Η νομοθεσία για τη θρησκεία αναφέρθηκε επίση. Εκπλήσωμε που από τι 300 τόσε θρησκείε μόνο 14 αναγνωρίζονται, αλλά και η ιδιοκτησία τους, γιατί άλλοι που δεν αναγνωρίζονται χάνουν και την ιδιοκτησία τους, από ό,τι φαίνεται οι άλλες θρησκείες. Τέλος, για το γάμο. Φυσικά, το οικογενειακό δίκαιο είναι εθνική αρμοδιότητα. Λέει, το να λέει στο Σύνταγμα ότι σε γάμο μπορούν ε, να πάνε μόνο ένας άντρας και μία γυναίκα, ε, αυτό είναι όπως και με τον νόμο για τον ε, τύπο, ότι δηλαδή ε, μπορεί να γίνεται έτσι διάκριση στα άτομα ομοφιλόφιλους, λεσβείες κλπ. Ευχαριστούμε Σόφη. Η Χάνστ. Ευχαριστώ. Θέλω να αναφερθώ σε τρία θέματα καταρχήν ε, στην ε, λεγόμενη πλειοψηφία. Οι πλειοψηφίες δεν έχουν πάντοτε δίκιο, έχουμε πολλά καλά παραδείγματα, ο καθένας μπορεί να κοιτάξει τη χώρα του και εμείς τη δικιά μας. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε πάντοτε ότι κάποιος έχει δημοκρατικά εκλεγεί και δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Διότι ε, αν υπάρχει εκλογή και τον του, της N5 ε, του κόμματος των εθνικοδημοκρατών στη Γερμανία ποιος μιλάει για δημοκρατία. Οπότε ε, πρέπει να κοιτάξουμε να προστατεύσουμε ό,τι είναι καλό από τις αρχές μας και να μην μιλάμε απλούστατα για να κάνουμε δηλώσεις. Ε, επίσης στα Δυτικά Βαλκάνια πολλές φορές λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και τώρα έχουμε το παράδειγμα της Ουγγαρίας όπου δεν συμβαίνει αυτό διότι η Ουγγαρία είναι στην οδό της πλήρους, ε, του πλήρους εκδημοκρατισμού και γι' αυτό σε αυτή την τελική ευθεία πρέπει να τους βοηθήσουμε και ε, το Κοινοβούλιο πρέπει να αντιδράσει ή να δράσει. Αυτό περιμένουν από εμά. Δηλαδή οι άνθρωποι που βγαίνουν στο δρόμο τώρα και διαδηλώνουν στην Ουγγαρία αυτό ζητούν, να συσπηρωθούν ως αντιπολίτευση και θεωρώ ότι είναι σημαντικό και έχω μόνο μία ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν να εμποδίσετε να δημιουργηθεί και πάλι ε, μία, ε, ε, ένα φιάσκο όπως στη Γαλλία όπου διαπιστώνουμε ότι αυτό το οποίο δεσμεύτηκε η Γαλλία να κάνει στο περίπτωση στο Ρωμά δεν έγινε. Δεν έγιναν πολλά πράγματα που έχουν δεσμευτεί να κάνουν και αν πρέπει να υπάρχει μία διαδικασία αθετήσεως στις συνθήκες ε, και αν η Επιτροπή λέγει ότι θα την εφαρμόσει πρέπει να υπάρξουν οι προποθέσεις τι ζητάμε λοιπόν ε, από την ε, Ουγγαρία η οποία θα μας απαντήσει όχι δεν υπάρχει ε, διαδικασία παρακάμψεως των συνθήκων. Τι θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή πώς θα, πώς πώς θα τους εμποδίσουμε να μην εφαρμόζουν τις συνθήκες. Ωραία. Και εγώ ζήτησα το λόγο και ζητώ την ε, Σόφη Ιντβέλτ να προεδρεύσει αν χρειαστεί. διότι και εγώ είμαι μέλος της Νομικής Επιτροπής της Ουγγαρίας και θέλω να σχολιάσω σχετικά με το τι γίνεται στην Ουγγαρία υπάρχουν κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές οι οποίες χρειαζόντουσαν και έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είτε δεν τις έπραξε ή δεν υπήρχε η πολιτική θέληση. Όλοι λοιπόν ήλπιζαν ότι θα υπάρξει αυτή η ρύθμιση διότι ε, αλλάξαμε τη, ε, ορισμένους νόμους. Όλοι ξέραμε ότι έπρεπε να γίνουν οι αλλαγές αυτές και ότι χρειάζονται οι, ε, αυτές οι αλλαγές. Οπότε υπάρχουν ορισμένα λάθη ε, τα οποία συμβαίνουν παντού και θα πρέπει ε, να δούμε εάν υπάρχει εφαρμογή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Υπάρχουν πολλά θέματα στα κράτη-μέλη τα οποία δεν ευθυγραμμίζονται με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και είναι πολύ σωστό ότι η Επιτροπή ε, εποπτεύει την εφαρμογή των συνθήκων και μπορεί να μας πει τι άλλαξε και αν υπάρχει ο σωστός μηχανισμός. Ας αφήσουμε λοιπόν την Επιτροπή να κάνει ό,τι χρειάζεται και δεν νομίζω ότι τα θέματα αυτά πρέπει να πολιτικοποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Για να επανέλθω σε αυτό που είπε η κυρία Λεμπάη, αν κοιτάξουμε όλα αυτά τα θέματα, ας δούμε τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχει μία ηλικία συνταξιοδοτήσεως η οποία διαφέρει 70 63 πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι οι δικαστές δεν μπορούν πλέον να εργαστούν αλλά όχι πλέον σαν δικαστές γιατί υπάρχει συνταγματικό όριο συνταξιοδοτήσεως και στη Γερμανία ξέρω ότι υπήρξε το θέμα αυτό, δηλαδή να υπάρχει όριο ηλικίες για ορισμένα επαγγέλματα. Έχουμε ε, επίσης την διαχείριση των δικαστηρίων η οποία αναλαμβάνεται από τα Υπουργεία. Ε, γιατί λοιπόν μας ενοχλεί διότι ε, είναι και αυτή ανεξάρτητη αρχή εφόσον έχει εκλεγεί μία αρχή από το Κοινοβούλιο είναι πιο ανεξάρτητη από ότι ε, η συνήθις. Υπάρχει καλύτερη εποπτεία, περισσότερες δυνάμεις και θα δείτε ότι παντού μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις και καλό θα ήταν να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτούς τους κανόνες. Ε, ξέρω ότι είναι δύσκολο να περιοριστώ. Μπορώ τώρα να συνεχίσω να προεδρεύω και έκλεισα τις παρατηρήσεις μου. Uh, I have Mrs. Alfano. Όλοι οι ομιλητές θα πάρουν το λόγο. Για να είμαστε ξεκάθαροι και να τηρήσουμε τον χρόνο θα σας πω. Then we have Mrs. Morvai, we have Mr. Foss, Mrs. Gomez, Mr. Michel, Mr. Alvaro, Mr. Mulder, Mr. Mulder. Yes. Mr. Sugar, Mrs. Boskurt and Mrs. Mr. Sire. Αυτά ήταν τα ονόματα στον κατάλογο μιλητών και κλείνω τον κατάλογο. Η κυρία Αλφάνο πρώτα. Εγώ συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπαν ήδη οι άλλοι συνάδελφοι, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω την Διευθύντρια Λεμπάη. Ε, ε, είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε και να ενεργούμε με, με ψηφίσματα, πράγμα που κάναμε ήδη. Ένα για, ψήφισμα εγκρίναμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ένα ε, για το Σύνταγμα. Εν τω μεταξύ όμως έκλεισε το Club Radio στην Ουγγαρία και χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτύρονταν και από αυτού εξέφρασε την άποψή της η Νέλη Κρούζ και εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες. Όπως έλεγε και η Σόφη, έγιναν αποδεκτές μόνο μόνο 14 ε, θρησκείες, ε, αποκλείοντας μάλιστα τη μουσουλμανική και τον βουδισμό. Έγινε η μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ στην απάντηση που δόθηκε στην Ουγγαρία. Όχι εκείνες οι πολύ μπανάλα απαντήσεις, ε, θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύετε εσείς εκεί που λέει η Ουγγαρία πως είναι απαραίτητο να υπάρχουν φιλόδοξοι και ευέλικτοι δικαστές. Τι θα πει δηλαδή ευέλικτος ε, δικαστής. Αδέκαστος πρέπει να είναι ο δικαστής ε, αμερόληπτος. Αυτός διαχειρίζεται τον νόμο προς το συμφέρον των πολιτών. Η ευελιξία τι σημαίνει εκεί. Ότι αν κάποιο είναι ισχυρό πρέπει να παριστάνει πως δεν τρέχει τίποτα και να κλείνει τα μάτια του. Αυτό είναι φρικτά πράγματα. Εγώ υποστηρίζω το αίτημα της ομάδας μου για την εφαρμογή του άρθρου 7 όχι απέναντι στην Ουγγαρία αλλά γιατί πρέπει να επιβεβαιωθεί και να γίνει σεβαστό το δικαίωμα, να είναι εγγυημένη ο σεβασμός της δημοκρατίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πάνω απ' όλα πρέπει να καταλάβουν 55 εκατομμύρια πολίτες και οι υπόλοιπε χώρες που μας παρακολουθούν ότι αυτά είναι θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά κυρίω από αυτού που ήδη είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα μ' άρεσε πολύ να πω μέλη των Ενωμένων Εθνών της Ένωσης, αλλά ίσως ποτέ δεν θα τα καταφέρουμε και κυρίως ίσως να μην έχουμε ποτέ συγκεκριμένα αιτήματα. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ε, ε, τους ε, αρχάριους σε σχέση με θέματα τα οποία ήδη θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Το μεταρρύθμιση των του δικαστικού σώματος είναι ad personam. Εγώ θα ήθελα να δω αυτούς τους δικαστές που είχαν 72, ε, που είναι 72 ετών και πάνω και που σίγουρα δεν βολεύουν πολύ τον Υπουργό και σίγουρα ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών στην Ουγγαρία. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εγγυηθούμε τον σεβασμό των συνθηκών της Ένωσης. Σας ευχαριστούμε κυρία Αλφάνο και κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ο Σουγκαρέζα, να ρωτήσω παρακαλώ κάτι την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα, ποιος, ε, ποιος κανόνας, ποιος νόμος του ευρωπαϊκού δικαίου εδώ αποτελεί και το λόγο, την αιτία για το γεγονός ότι εντοπίζονται παραβιάσεις. Το 2006 στην Ουγγαρία υπήρξαν φασαρίες, παραβιάσεις, είχαν ε, διωχτεί εκατοντάδες και είχαν απειληθεί από την αστυνομία ένας οροκόσμος. Τώρα λοιπόν θέλω να ξέρω ποια είναι η νομική βάση που το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξεκίνησε τη διαδικασία βάση του άρθρου 7 και δεν αντέδρασε καθόλου τότε σε αυτές τις μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποια είναι η νομική βάση για αυτή την έλλειψη δράσης. Πέρα το ότι εγώ η ίδια ήμουν παρούσα στις παραβιάσεις αυτές και είμαι και δικηγόρος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και δουλεύω με τα θύματα, Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να παραμείνω ήρεμη σε μια τέτοια ανταλλαγή απόψεων όπως αυτή που έχουμε σήμερα. Γι' αυτό και θα διαβάσω τα υπόλοιπα, ώστε να μην ε, με πιάνει ο ενθουσιασμός. Η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αυτό που διέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και το πρώτο άρθρο λέει τα εξή. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα αυτοδιάθεση. Παραβίαση τέτοιου δικαιώματο δεν μπορεί να υπάρχει. Πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν να ακολουθούν τα πολιτικά τους ε, συστήματα και να φροντίζουν για την οικονομική τους ανάπτυξη. Είναι πολύ βασικό αυτό συλλογικό δικαίωμα. Είναι αρχή διεθνούς δικαίου, είναι νομοθεσία η οποία ισχύει και υπάρχει σε όλες τις χώρες. Κάθε λαός έχει δικαίωμα το κράτος του. Έτσι λέει το νομοθετικό αυτό κείμενο. Και υπάρχει ένα δικαίωμα για όλους τους λαούς σε αυτοδιάθεση. Άρα και οι Ούγγροι έχουν αυτό το δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Ο Ουγγρικός λαός δεν μπορεί να χάσει αυτό το δικαίωμα. Δεν μπορεί να χαρίσει το κράτος ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε στις τράπεζες, ούτε σε κανέναν. Δεν μπορεί να πουλήσει το δικό του θεμελιώδες δικαίωμα ο λαός της Ουγγαρίας με κανένα αντάλλαγμα. Το Ουγγρικό κράτος δεν μπορεί να παραχωρήσει το δικαίωμα αυτό που έχει ο λαός του σε κανέναν, γιατί είναι δικαίωμα του λαού. Η συζήτηση που κάνουμε σήμερα έχει ως τίτλο «Κατάσταση στην Ουγγαρία». Ξεχνάτε όμως αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα. Όλη η νομοθεσία είναι νομοθεσία η οποία έχει να κάνει με την αυτοδιάθεση του λαού. Υπάρχει πρόβλημα στην Ουγγαρία. Ναι, πολλά προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, αλλά όχι αυτά που νομίζετε εσείς, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε άλλοι εκπρόσωποι αν υπάρχει κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό είναι γιατί οι Ουγγροί ζουν σε μεγάλη φτώχεια, γιατί υπάρχει μεγάλη ανεργία. Ακόμα και αν έχουν διπλώματα, πολλοί αναγκάζονται να δουλεύουν σε πολύ κατώτερων προσόντων ε, απασχόληση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι πράγματα τα οποία δεν είναι συμβατά με αυτή την κατάσταση που ζουν οι Ούγγροι. Και μάλιστα ε, δουλεύουν και με επικίνδυνη εργασία. Το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Εγώ το λέω και στους συναδέλφους από την ΚΟΕ, ότι το δικαιώματα στικαλιστικά δεν υπάρχουν. Πολλοί γεωργοί δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Ή αν το κάνουν, τα πουλάνε σε πολύ χαμηλές τιμές που δεν ανταποκρίνονται ούτε καν στο κόστος. Και πολλοί άνθρωποι δουλεύουν για 300 ευρώ το μήνα. Ναι, ναι, και μην με σταματάτε, ναι, ναι. Μην μου κόβετε το λόγο. Θέλουμε να υποστηρίξουμε το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση. Οπότε αφήστε με, κυρία Πρόεδρε. Αν μου κόψετε το λόγο, κυρία Πρόεδρε, εγώ θα πρέπει να βρω άλλο τρόπο για να μ' ακούσετε και να μ' ακούσουν οι συνάδελφοι. Εγώ θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στις ερωτήσεις μου. Διακόπτη, Πρόεδρος. Θέλω να υποστηρίξω τους Ευρωπαίους εργαζόμενους, λέμε Λιτρία. Ήμουνα πάρα πολύ γενόδορη μαζί σας, λέει η Πρόεδρος. Σας έδωσα τα πέντε λεπτά. Και εντάξει, το ζήτησε ο κύριος Κλέης, το έκανα. Ως εκεί. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Φόξ έχει το Ευχαριστώ. Αυτό που ακούω εγώ είναι εδώ πολιτικά ευχολόγια σαν βάση συνεργασίας και συμβιώσεως και αντιλαμβάνομαι ότι ουσιαστικά πρέπει να συμβιώνουμε βάση του δικαίου, διότι διαφορετικά θα υπάρχει αυθαιρεσία ενδεχομένως χρειάζονται ορισμένες αλλαγές ακόμη και στο νόμο του τύπου αλλά ε, εφόσον ε, είναι αποδεκτά πρέπει να τα αποδεχόμαστε κάποια στιγμή και το μέτρο του ελέγχου αυτού πρέπει να είναι ε, το, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και καταλαβαίνω την κυρία Ντεμπάη ότι εάν η κατηγορίες προσκρούν ή στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που πρέπει να θεωρηθεί σαν το ισχύον μέτρο, τότε θα πρέπει να στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχήν και όχι υποχρεωτικά στα κράτη-μέλη ε, διότι ε, ε, νομικά υπάρχουν δυσκολίες μπορεί να δικαιολογούνται πολιτικά ή ηθικά διότι τότε αν υπάρχουν βάσει των θεμελιωδών δικαιωμάτων δημεύσεις περιουσιών 100 χιλιάδων ατόμων, τότε αν αυτό προβλέπεται από το χάρτη θα πρέπει να καλύπτεται. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι εδώ υπάρχει μία συνήθις διαδικασία παραβιάσεως των συνθήκων ε, και ε, τι γίνεται σε άλλες χώρες όταν δεν ε, υπάρχει αυτή η διαδικασία και ο χρόνος για να τα συζητήσουμε. Για μένα είναι μια φυσιολογική διαδικασία παραβίασης των συνθήκων και πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά πρέπει να διαπιστώσουμε ότι το μέτρο και σταθμό πρέπει να είναι ε, εδώ ένα και έχω εμπιστοσύνη στην Επιτροπή ε, και τη ρωτώ υπάρχει παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ναι ή όχι διότι η βάση της συμβιώσεώς μας πρέπει να παραμείνει ε, το δίκαιο και πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόζουμε το δίκαιο μέσα στα μέτρα του δυνατού και άρα αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την τελευταία φορά που βρισκόμουν στην Ουγγαρία παρακολούθησα μια ε, πολύ ωραία, έναν ωραίο εορτασμό, μια τελετή ε, στο, Ευρω... στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Μετά βγήκα έξω, είδα μια αμερικανική αντιπροσωπεία διπλωματών μαζί με Ευρωπαίους διπλωμάτες. Ήταν μια ομάδα, βεβαίως ήταν μεγάλη παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τους ρωτήσαμε τι συμβαίνει και πρέπει να σας πω προς λύπη μου πως όλοι τους αυτοί που ζούσαν στη Βουδαπέστη μας ε, έδωσαν την εντύπωση μας ε, ότι πρόκειται για ένα πολύ αυταρχικό, φασιστικό καθεστώς. Εγώ τρόμαξα. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησαν όμως. Αλλά όταν είδα τι συμβαίνει, γιατί όσον αφορά το νόμο περί μέσων μαζική ενημέρωση, τίποτα δεν βελτιώθηκε έκτοτε. Αντίθετα, κλείσαν ένα σωρό σταθμοί, ένα εκατοντάδες επαγγελματίες έχουν φύγει, έχουν ε, μάλλον απολυθεί ε, και επικρατεί λογοκρισία, γίνεται λογοκρισία και μετά είδαμε την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας για το νέο σύνταγμα. Εξετάσαμε, εξετάζουμε το εκλογικό νόμο. Σύμφωνα με αυτό τον εκλογικό νόμο υπάρχει υπάρχει δυνατότητα το κεντρικό κόμμα τη αντιπολίτευσης να θεωρηθεί παράνομο. Είδαμε όλα τα στοιχεία που ανέφερε η κυρία Λεμπάη, η ε, ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, προστασία δεδομένων, Εθνική Τράπεζα κτλ. Μα είναι μια ολόκληρη εικόνα, δεν είναι μόνο η Ουγγαρία. Είναι, αφορά εμάς, την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά εμένα, εμένα προσωπικά, την Πορτογαλία, το είδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία είμαστε μέλη. Ε, αυτοί οι οποίοι έπρεπε να είναι θεματοφύλακες στις συνθήκες δεν έκαναν τη δουλειά τους. Ε, λυπούμε που σας το λέω, είμαστε σήμερα εδώ γιατί η Κομισιόν δεν έκανε τη δουλειά της και ούτε το Συμβούλιο έκανε τη δουλειά του. Και είναι σωστό λοιπόν το Κοινοβούλιο να κάνει τη δική του δουλειά και να τους πιέσει να κάνουν αυτό που είναι απαραίτητο. Και πρέπει να πω ότι αυτό δεν είναι, γίνεται κατά του γκρικού λαού, αλλά υπέρ του γκρικού λαού λαού καθώς και υπέρ όλων των λαών μας γιατί ζούμε σε αυτή την κοινή Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή είμαστε μια κοινωνία που σέβεται τον νόμο και τα δικαιώματα. Ευχαριστούμε. Κύριε Γκόμες, δεν μου κάνετε πολύ εύκολο το έργο μου ως Προέδρου. Ο κύριος Μίτσελ τώρα έχει το λόγο. Ο κύριος ε, Λουί Μισελ, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, Κυρία Πρόεδρε, κυρία Γενική Διευθύντρια, ο τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση, εμένα με προβληματίζει. Βλέπω ότι διάφοροι είναι σε αποστολή, κύριε Έγγελς. Καταλαβαίνω και εσείς, κύριε Γκάλη, ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Οπότε, κύριε Έγγελ, να ξέρετε ότι αυτά που θα πω εγώ δεν θα είναι ιστερικά, δεν θα είναι ιστερική η παρέμβασή μου. Απλώς πρόκειται για το θεμελιώδες δικαίωμά μου ως Ευρωβουλευτού. Και εξάλλου ούτε αισθάνομαι ότι οι ερωτήσεις μου και τα σχόλιά μου ε, περνάνε από ένα λαϊκό δικαστήριο. Θα ήταν τρομερό να θεωρήσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν πολυφρόνημα ε, φροντίζει να τίθεται σε εφαρμογή τα δικαιώματά του είναι σαν να πρόκειται για λαϊκό δικαστήριο. Όχι, αλλά όλες αυτές οι αξίες είναι αξίες ευρωπαϊκές που είπαμε. Φυσικά έχω ακούσει και κάτι τερατώδες. Μπορεί να πέρασε στα ψηλά, αλλά η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι στα κράτη-μέλη, άκουσα. Μα τι τερατώδες είναι αυτό. Τερατώδες. Αυτοί που σήμερα κάπως απλοποιούν τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ουγγαρία είναι έτοιμοι να καταδικάσουν ε, παραβιάσεις όταν αυτές γίνονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα εγώ νομίζω ότι είναι θέμα ηθικής. Όταν τέτοιες παραβιάσεις γίνονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε χρέος να τις καταγγέλουμε. Είτε με καθυστερήσεις, είτε κοφεύοντας, με τη συνενοχή ακόμα θα έλεγα πολλές φορές. Έτσι οδηγούμαστε σε μια βαθιά κρίση αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης και χάνει το νόημά του το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Εδώ πρέπει να σας το πω έντονα, συνάδελφοι. Όχι, δεν είναι χωρίς σημασία. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Όχι, είναι τρομερό η ίδια αυτή η ιδέα για την Ευρώπη που είναι ανθρωπισμός, που είναι άνοιγμα, που είναι αλληλεγγύη, που είναι πρόοδος, που είναι δικαιοσύνη, η ισότητα. Με δύο λόγια, οι οικουμενικές αξίες και είναι και η απόρριψη καθενός που προσπαθεί να μεροληπτήσει. Πρέπει να βλέπουμε τις πράξεις. Και αυτό ακριβώς που εγώ λέω είναι ότι λείπει και είναι μεγάλο αμάρτημα αυτό που κάνουμε το να μεροληπτούμε δηλαδή να βάζουμε μια χώρα στην υπηρεσία μιας πολιτικής δύναμης. Έχετε πρόβλημα κυρία Πρόεδρε, ποιο είναι το πρόβλημά σας. Δεν αισθάνεστε άνετα, ε? Το καταλαβαίνω αυτό ότι δεν αισθάνεστε άνετα, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι τα μέτρα αυτά, υπενθυμίζω, τα μέτρα αυτά είναι πράξεις, δεν είναι προθέσεις. Και όταν αυτά τα συγκρίνει... Κύριε Μισελ, θα σας αφαιρέσω το λόγο γιατί έχετε περάσει το χρόνο το οποίο σας έχω διαθέσει. Αυτό σας έλεγα. Δεν σας κατάλαβα. Θα συνεχίσω και θα συνεχίσω να ουρλιάζω αν μου κόψετε το μικρόφωνο. Όχι, ουγγρικά δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, εντάξει, θα τελειώσω γρήγορα. Θα είμαι σύντομος. Λίγα πραγματάκια έχω ακόμα να σας μεταφέρω. Λοιπόν, τι γίνεται στην Ουγγαρία σήμερα, σε μια χώρα δηλαδή ευρωπαϊκή. Αυτό που γίνεται είναι μια μετάλλαξη ουσιαστικά. Κόβει το λόγο η πρόεδρος. Είχαμε και την κυρία Βίμπερ, η οποία για πέντε λεπτά εκ μέρους της ομάδας σας πήρε το λόγο. Τώρα οι υπόλοιποι έχετε λιγότερο χρόνο. Είχα πει δύο με τρία λεπτά. Ήμουν ήδη αρκετά γενναιόδορη μαζί σας κύριε Μισελ, οπότε σας αφαιρώ το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Μισελ. επόμενο στον κατάλογο μιλητών είναι ο κύριο Άλβαρο. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε σε αυτό το σημείο μπορώ να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Λουί Μισελ με τον ίδιο ενθουσιασμό και με τις ίδιες ανησυχίες. Το θέμα δεν είναι μόνο η Ουγγαρία και το έχουμε πει αρκετές φορές. Δηλαδή όταν υπάρχει μία τέτοια συμπεριφορά ενός κράτους μέλους είτε πρόκειται για τη Γερμανία είτε την Ουγγαρία είτε τη Μεγάλη Βρετανία και ανέφερα μόνο λίγες δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα διότι πρέπει να σας πω ότι σε θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων η πλειοψηφία των κρατών ε, ε, έχει κάνει μουσκεμα ε, και συμπεριφερόμαστε χειρότερα ίσως από τα μη κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες θα άξιζαν ορισμένες επιπλήξεις ή απειλές για να διορθώσουν την εσωτερική τους κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να φωνάζουμε περισσότερο για τις τρίτες χώρες από ότι ε, μέσα στην οικογένειά μας και να μην υπάρχει πειθαρχία. Θα έπρεπε να κανονίσουμε τα του, και να ρυθμίσουμε τα του οίκου μας και μετά τον έξω. Και αυτό δεν αναφέρεται ή σε την συμμετοχή ενός κράτους μέλους διότι θα ήταν ε, κακό μέτρο να χρησιμοποιήσουμε κάτι τέτοιο ούτε μπορούμε να ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές διότι αν υπάρχει απειθαρχία στις αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες που θα κάνουν τα ίδια και νομίζω ότι το Συμβούλιο δεν έχει δίκιο αν αφήνει ε, την ε, Επιτροπή σαν μοναδικό θεματοφύλακα των συνθήκων και την αφήνει να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει την αρμόζουσα διαδικασία και θα πρέπει να δούμε βάσει ποιων κριτηρίων. Δηλαδή το άρθρο 7 μπορεί να ισχύσει βάσει του άρθρου 2. Πρέπει να δούμε ε, τι ε, θέμα υπάρχει με την ανεξαρτησία της ε, κεντρικής τράπεζας ε, του τύπου των δικαστών διότι νομίζω ότι αυτά είναι θέματα της συνθήκης της Λισαβόνας η οποία αναπτύσσεται σε όλα αυτά τα σημεία και δεσμεύει όλα τα κράτη σε ό,τι διατυπώνεται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν θέλω να να με αποπέμψετε και γι' αυτό θα πω ακόμη ένα θέμα αγαπητή Κίνγκα όντως ήταν λάθος αλλά τα λάθη υπάρχουν για να διορθώνονται και έτσι που βλέπουμε να επαναλαμβάνονται τα λάθη αυτά θα καταλήξουν σε μία παραπομπή και τότε δεν πρόκειται για λάθος πρόκειται ε, για δόλια κίνηση και τελικά τελειώνω λέγοντας ε, ότι αυτό ισχύει και για την Επιτροπή και για το Συμβούλιο και για όλους. Είναι κανείς υπέτειος όχι μόνο όταν λειτουργεί αλλά όταν δεν αναλαμβάνει δράση. Και ο κύριος Σόμπερ είναι τελευταίος. Σας ευχαριστώ. Εγώ μιλώ ως απλό μέλος και όχι ως ε, δεύτερος συντονιστής του ΕΛΚΑ. Κίνγκα, ανέφερε ήδη τι πρώτε μου παρατηρήσει και δεν χρειάζεται να τι επαναλάβω σε σχέση με την ανεξαρτηστή ε, διοίκηση των δικαστηρίων. Όμω, δύο συναδελφοί μου μίλησαν για τον νόμο περί εκκλησίας και περί των ε, ραδιοφωνικών σταθμών. Θα πρέπει να πω πω το Συμβούλιο Μέσων Μαζική Ενημέρωση δεν έχει αποσύρει την ε, συχνότητα του Club Radio, ούτε το έχει αναγκάσει να κλείσει. Μπορώ να σα δώσω τι λεπτομέρειε, χρειάζεται να χασομερίσω με αυτό. Ξέρω μόνο για ένα ραδιόφωνο, ένα ραδιοφωνικό σταθμό που απαγορεύθηκε στη Σλοβακία ε, λόγω του σλοβακικού νόμου περί γλώσσας και μάλιστα ήταν ένας αγγλόφωνος σταθμός. Τώρα, στα 27 κράτη-μέλη υπάρχουν 5 ε, ή μάλλον 9 κράτη-μέλη ε, για πέρα από την Ουγγαρία, όπου λιγότερες από 14 εκκλησίες αναγνωρίζονται. Στο Βέλγιο μόλις 6 εκκλησίες αναγνωρίζονται. Και οι αναγνωρισμένες 14 εκκλησίες αντιπροσωπεύουν το 99% του ουγγρικού πληθυσμού. Και αν προχωρήσουμε περισσότερο και εξετάσουμε τον νόμο περί εκκλησιών, υπάρχουν άλλες εκκλησίες που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για καταγραφή και ήδη 83 έχουν ζητήσει να καταγραφούν. Κάτι ακόμα. Εάν συγκρίνουμε με πολλά άλλα κράτη-μέλη, στην Ουγγαρία δεν υπάρχει εθνική θρησκεία, αναγνωρισμένη θρησκεία του κράτους. Σε άλλα κράτη υπάρχει αυτό, στην Ουγγαρία όχι. Αυτά λοιπόν περί του νόμου για την ε, Εκκλησία και ως μέλος Ευρωβουλευτής ε, θα πρέπει να αρνηθώ και θα θέλω να διαμαρτυρηθώ για τέτοιες κα, κατηγορίες που ανέφεραν οι συνάδελφοι ότι στην Ουγγαρία υπάρχει κυβέρνηση, ατμόσφαιρα που δείχνει πως υπάρχει επικρατή επικρατεί φασισμός στη χώρα αυτή τότε εγώ θα έλεγα ότι εφόσον προέρχομαι από μια πρώην κομμουνιστική χώρα θα έπρεπε να πω ότι όλοι μου οι σοσιαλιστές, οι σοσιαλιστές συνάδελφοι είναι σταλινιστές. Θα έπρεπε έτσι να τους αποκαλώ όλους. Όχι, ε, διαμαρτύρομαι και πρόεδρε και εσείς θα πρέπει να διαμαρτυρηθείτε αν κάποιος λέει πως... Ε, ισχύει κάτι τέτοιο στην Ουγγαρία. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε, αλλά επαναλαμβάνω άλλη μια φορά πως ο ραδιοφωνικό σταθμό δεν έκλεισε στην Ουγγαρία. Κοιτάξτε λίγο καλύτερα τι συνέβη με αυτό το σταθμό, το Club Radio και θα καταλάβετε. Και μην πιστεύετε όσα λέει ο τύπο στι εφημερίδε. Ευχαριστούμε κύριε Σόγκορ. Μόλτερ. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Μούλτερ. Δεν είναι η πρώτη, φορά. που συζητάμε για την Ουγγαρία. Το έχουμε κάνει και κατά το παρελθόν και υπό Ουγγρικής Προεδρίας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, τι είναι αυτό που θα κάνει τελικά την Επιτροπή να προχωρήσει αντί να κάθεται να μελετάει. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 10 μιλάει για ελευθερία συνείδησης και θρησκείας. Όλοι έχουν αυτό το δικαίωμα που σημαίνει και την ελευθερία να αλλάξει κανείς θρησκεία κλπ. κλπ. Δεν λέει ότι πρέπει να έχετε ένα συγκεκριμένο αριθμό εκκλησιών, όπως λέμε τώρα για την Ουγγαρία. Για μένα αυτή είναι παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Θα μπορούσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει είναι αλήθεια ότι στις 17 Ιανουαρίου θα αποφασίσουν να πάνε στο δικαστήριο, ναι ή όχι. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να έχουμε επιτέλους μια ανεξάρτητη αρχή η οποία κρίνει γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μόνη της δεν φαίνεται να τα καταφέρνει. Η κυρία Μπόσκοτ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, έχω και εγώ να ρωτήσω κάτι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν είναι η πρώτη φορά που μας λέει για την Ουγγαρία και σήμερα έχει να κάνει με το Σύνταγμα της ε, Ουγγαρίας και για τις θεμελιώδεις αξίες σωστά κοιτάει να δει τι είναι αυτό το οποίο δεν είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο εφόσον η Ουγγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Όμως τα συζητήσαμε αυτά και όταν είχαμε να κάνουμε με το νόμο για τον τύπο. Δεν φαίνεται ότι κάναμε αυτό που έπρεπε. Ο, η Ρέντινγκ που είναι αρμόδια δεν ασχολήθηκε με το τεχνικό επίπεδο, με τις τεχνικές λεπτομέρειες του νόμου και τελικά έχω την εντύπωση ότι η Επιτροπή έχασε μια ευκαιρία. Ρωτάω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, πόσε πιθανότητε υπάρχουν να γίνει το ίδιο και αυτή τη φορά. Μήπω θα έπρεπε με κάποιον άλλο τρόπο να χειριστεί το θέμα για να μην αποτελέσει όλη αυτή η διαδικασία ένα κακό παράδειγμα και για άλλες χώρες. Μήπως θα έπρεπε να κοιτάξετε καλύτερα τι διαδικασία θα ακολουθήσετε αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Μπόσκορτ. Ο κύριος Σάγια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πώς ορίζω εγώ το φασισμό ή τον ε, κομμουνισμό, δεν είναι τίποτα άλλο από το να ε, καταδικάζεις ε, μεταξύ τερού και αχλαδίου χωρίς καμία πραγματική έρευνα. Έχοντας ακούσει λοιπόν τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ, θέλω να απορρίψω αυτά που είπε η κυρία Κόμες για την Ουγγαρία, ότι είναι φασιστική κλπ. Ποτέ δεν πρέπει κανείς να κρίνει πριν ε, γίνει η δίκη. Είναι κάτι που το ζήσαμε κι εμείς. Το λέω λοιπόν και εδώ στο Κοινοβούλιο προσοχή, πριν καταλήξετε συμπεράσματα, ερευνήστε πρώτα. Και όπως άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώς αυτό ξεκαθάρισαν. Και νομίζω ότι είναι σωστό. Στην Ουγγαρία, τον τελευταίο χρόνο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είχαμε ένα νέο σύνταγμα. Ακούστηκαν επικρίσεις ότι μέσα σε νέα μήνες πέρασε. Σας υπενθυμίζω ότι η νέα συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζητάμε τώρα σε 4, 5 ή 6 εβδομάδες θα τεθεί σε ισχύ, που είναι επίση ένα πολύ σημαντικό έγγραφο. Επίσης, πέρασε με 200, πέρασαν 230 νόμοι από το Κοινοβούλιο και η χώρα μετά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και την κυβέρνησή του ήταν υποκατέρευση, δεν υπήρχε ασφάλεια, ε, ξέρετε όταν έφυγε ο από την ε, κυβέρνηση, τι έγινε με τον προπολογισμό, με το χρέος. Πραγματική καταστροφή. Οι δημόσιες υπηρεσίες ήταν υποκατάρρευση. Το είπατε κι εσείς ότι στους δρόμους κυκλοφορούσαν ε, παραστρατιωτικές δυνάμεις, γιατί η αστυνομία, η κυβέρνηση δεν μπορούσαν να προσφέρουν ασφάλεια στους πολίτες. Εγώ είμαι από το Φιντές, να ξέρετε, για όσους δεν το γνωρίζουν. Εμείς Λοιπόν, από το Φιντες τι κάναμε, κληρονομήσαμε μια τέτοια κατάσταση. Που και εμείς βγήκαμε στην εξουσία επειδή ακριβώς ο κόσμος ήθελε αλλαγή. Όχι γιατί τραβήξαμε τον πρώτο λαχνό. Και αν περάσαμε αυτούς τους νόμους είναι γιατί ακριβώς θέλουμε τη δημιουργία μιας νέας χώρας που να λειτουργεί. Να κοιτάξουμε λοιπόν από πίσω γιατί έγιναν όλα αυτά. Αυτό ήταν ο λόγο. Αν έγιναν μόνο 4-5 λάθη σαν και αυτά που εντοπίζετε εσεί εδώ, ε, είμαι πολύ ικανοποιημένο. Γιατί μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα πώ θα γινόταν αλλιώ. Αν μόνο 4-5 ή 6 σημεία είναι αυτά τα οποία σα ε, ανησυχούν, εγώ θα είμαι ευχαριστημένο. Πιστεύω ότι το, Ευρωπαϊκό... το Ουγγρικό Κοινοβούλιο έκανε πολύ καλή δουλειά με του νόμου που ενέκρινε. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να το ερευνήσετε πράγματι και συμφωνώ με αυτού που λένε ότι το Κοινοβούλιο είναι αυτόνομο και έχει το δικό του δικαίωμα να ασχοληθεί με την υπόθεση. Αλλά σκεφτείτε, όλη αυτή η νομοθεσία που το 90% δεν έχει ακόμα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες και ακόμα ε, με τις μεταφράσεις φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνετε το νομικό σύστημα που υπάρχει από πίσω, τη διασύνδεση μεταξύ τους. Πρέπει να καταλάβετε ότι είναι τεράστια ευθύνη για το Κοινοβούλιο να πάρει μια απόφαση. Το, η Κομισιόν μπορεί να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξει σε αυτήν την απόφαση. Ευχαριστώ λοιπόν και να πω στους συναδέλφους που κατέκριναν την Ουγγαρία ότι δεν ακολουθεί τους ευρωπαϊκούς νόμους. Μα κύριε Μισελ, αν εσείς δεν μπορείτε να τηρήσετε τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε εδώ σε αυτή τη συνεδρία για το πόσο χρόνο μιλάει κανείς, πώς μπορείτε να πετήσετε από την Ουγγαρία να τηρεί. Ε, αναφέρθηκε σε μένα. Ο κύριος θέλω να το απαντήσω. Α, όχι, όχι, όχι, έχω δικαίωμα ε, να απαντήσω. Λοιπόν, θέλω να επενθυμίσω, αγαπητέ συνάδελφε, ότι είναι δικαίωμά μου, απόλυτο δικαίωμά μου, να τοποθετούμε όχι απέναντι σε προθέσεις, όχι απέναντι σε κάποιο πρόγραμμα, να τοποθετούμε απέναντι σε πράξεις. Είναι δικαίωμα κάθε ευρωβουλευτή να το κάνει. Αλλά δεν υπάρχει καμιά αφιβολία ότι εσείς συνηθίζετε να μην τηρείτε το κοινοβουλευτικό κανόνα. Πρόεδρος, σταματήστε, σας αφαιρώ σε όλους το λόγο. Η κυρία Λεμπάιλ τώρα θα προσπαθήσει να απαντήσει στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Παρακαλώ κυρία Λεμπάιλ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω λεπτομερώς όλες αυτές τις ερωτήσεις που μου υποβάλλατε. Αυτό που θα προσπαθήσω λοιπόν να κάνω είναι να συγκεντρώσω ε, τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν αναθέματα. Το πρώτο θέμα λοιπόν που αναφέρθηκε από διάφορους ευρωβουλευτές είναι το τι συμβαίνει και κατά πόσο όταν υπάρχει μια υποψήφια χώρα τυχαίνει διαφορετικής μεταχείρισης από ό,τι χώρες μέλη δεν υπάρχει αυτή η διάκριση δηλαδή ανάμεσα σε υποψήφιες και χώρες μέλη. Κοιτάξτε, από τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα, το γεγονό ότι την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια και πάλι θα συζητηθεί αυτό, το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένα από τα μέσα της προηγούμενης χρονιάς και ξανά το Δεκέμβριο όταν ήταν σαφές ότι οι νόμοι αυτοί γινόντουσαν πιο συγκεκριμένοι, παρενέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ξεκάθαρα ότι καμία χώρα μέλος δεν μπορούσε να παραβιάζει τις συνθήκες ή τη χάρτα θεμελιδών δικαιωμάτων. Και η, και η δουλειά που κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ακριβώ αυτό, να διασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη απάντηση και είναι κάτι που ισχύει για τις χώρες μέλη αλλά και τις υποψήφιες χώρες. Αυτά τα βλέπετε και στην δήλωση που έκανε αντιπρόεδρος Ρέντινγκ στην Ολομέλεια τον Ιούνιο που μας πέρασε, όταν είπε ότι τα κράτη-μέλη έχουν κάθε δικαίωμα να τροποποιούν το σύνταγμά του να υιοθετούν νέο σύνταγμα, αλλά επίση, ξεκαθάρισε ότι το σύνταγμα αυτό θα πρέπει να συνάδει με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, κανόνες και με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Υπό το πνεύμα αυτό λοιπόν εμείς εργαζόμαστε. Και δεν βλέπω να γίνεται καμία διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτό που προσπαθεί να πετύχει το Κοινοβούλιο και αυτό που προσπαθεί να πετύχει η Επιτροπή. Βέβαια το κάθε θεσμικό όργανο έχει το δικό του ρόλο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακα των συνθήκων έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο και μπορεί να δράσει μόνο βάσει μιας ε, πολύ δυνατής πολιτικής ανάλυσης και νομικής μάλλον, νομικής ανάλυσης. Εφόσον από 1η Ιανουαρίου έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται οι νέοι αυτοί οι νόμοι και σήμερα πώς έχουμε, 12 Ιανουαρίου, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ήδη από το Δεκέμβριο να δουλεύει εντατικά πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα περίπλοκα. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε σε έννοιες όπως είναι η επανένωση οικογενειών. Εδώ πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα νομικά στοιχεία βάσει των οποίων να αποφασίσουμε, τα οποία να είναι αδιαμφισβήτητα από νομική άποψη. Επίσης, Όλοι δεχόμαστε ότι δεν πρόκειται για ένα καθαρά νομικό ζήτημα, ότι πρόκειται και για νομικό αλλά και για πολιτικό ζήτημα. Συνεπώς, έρχομαι έτσι στο δεύτερο θέμα. Ποια είναι η νομική βάση, ρωτάτε, πάνω στην οποία δουλεύουμε για να ελέγξουμε το κατά πόσο συμμορφώνονται οι ουγγρικοί νόμοι με το κοινοτικό δίκαιο. Η απάντηση είναι πολύ απλή όσον αφορά τη συνταξιοδότηση των δικαστών, την ηλικία τους δηλαδή, κοιτάμε κατά πόσο είναι συμβατή η ρύθμιση αυτή με την οδηγία 278 που αναφέρεται στη μη διάκριση όσον αφορά την απασχόληση. Για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης κοιτάμε το συμβατό με το άρθρο 47 της χάρτας που βέβαια συνδέεται άμεσα με το άρθρο 2 της συνθήκης. Και όσον αφορά την ανεξαρτησία του επόπτη της αρχής προστασίας δεδομένων, εδώ κοιτάμε κατά πόσο συνάδει με την οδηγία για την προστασία δεδομένων του 95. Αυτό ήταν το δεύτερο θέμα, λοιπόν, στο οποίο αναφερθήκατε. Υπήρξε και μια τρίτη κατηγορία ερωτήσεων που ήταν τελικά τι περιμένετε από την Ουγγαρία. Αυτό που εμείς προσδοκάμε από την ε, Ουγγαρία ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα είναι πλήρη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο. Πλήρη συμμόρφωση με το γράμμα και το πνεύμα των συνθήκων και τη Χάρτα Θεμελιδών Δικαιωμάτων. υπήρξε και ένα ερώτημα που ήταν τι θα κάνει την επόμενη εβδομάδα, τι θα αποφασίσει η Κομισιόν την επόμενη εβδομάδα. Ε, δεν μπορώ να σας πω τι θα αποφασίσει την επόμενη εβδομάδα η Κομισιόν, γιατί η Κομισιόν θα αποφασίσει βάσει της ανάλυσης που θα έχει στη διάθεσή της. Και εννοείται ότι είναι δικαίωμα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποφασίσει αυτό που κρίνει ορθό τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό πάντως που μέχρι τώρα έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να εκφράσει βαθιά ανησυχία με τον πρόεδρο και τρεις αντιπροέδρους που έστειλαν επιστολή στις Ουγγρικές Αρχές και βάσει της νομικής ανάλυσης που θα έχουμε στη διάθεσή μας σε χρόνο ρεκόρ, έτσι, την επόμενη εβδομάδα, είπαμε 17 Ιανουαρίου, θα είναι έτοιμα ε, και οι νόμοι αυτά να εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, σε χρόνο ρεκόρ θα πάρει την απόφασή τη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποιώντα πλήρω τα δικαιώματά τη ω θεματοφύλακα τη συνθήκη. Και το ξέρετε κι εσεί, κύριε Μέλντερ, αυτό είναι ο ρόλο τη. Και βάσει αυτού του ρόλου μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο και να πάει κάποια χώρα μέλο στο δικαστήριο επί παραβάση. Αλλά θα τα ξέρουμε όλα αυτά την επόμενη εβδομάδα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντεμπάιλ και για το χρόνο που μας διαθέσατε. Έχουμε καθυστερήσει 30 λεπτά σε σχέση με την ημερήσια διάταξη, οπότε κλείνουμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη και περνάμε ευθύς αμέσως στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα το απόγευμα. Αυτό είναι το πολιτέ πλαίσιο για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωση για την περίοδο 2013-2017. Λίγα λεπτά θα διακόψουμε μέχρι να αποχωρήσετε από την αίθουσα, όσοι θέλετε.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 Παρακαλώ, καθίστε για να εξετάσουμε το τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης. Πρόκειται για το πολιτές πλαίσιο για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2013 μέχρι 2017. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 168 για την δημιουργία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, οι θεματικοί τομείς των δραστηριοτήτων θα οριστούν μέσω ενός πενταετούς πολιετούς πλαισίου. Το ισχύον πλαίσιο εκπνέει στο τέλος του 2012 και η υιοθέτηση αυτής της, στόχος αυτής της πρότασης είναι να δημιουργηθεί ένα πολιετές πλαίσιο για αυτόν τον οργανισμό για την περίοδο 2013 μέχρι 2017 όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του κανονισμού. Επειδή δεν έχουμε εισηγητή, θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν για να μας παρουσιάσει λεπτομερώς την πρότασή της και βεβαίως αν κάποιος συνάδελφος θέλει να παρέμβει θα μπορέσει στη συνέχεια και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα όταν θα έχουμε ορίσει εισηγητή. Δίνω τώρα το λόγο στην Επιτροπή για να μας παρουσιάσει την πρότασή της με λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήδη θυμήσατε το πλαίσιο. Έχετε λοιπόν ενώπιόν σας μια πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την δημιουργία ενός πολιετές τους πλαισίου που θα καλύψει τα έτη 2013 μέχρι 2017. Όπως είπατε, πρόκειται για μία απέτηση του κανονισμού δημιουργίας του οργανισμού είναι για τον ορισμό ενός πολιτούς πλαισίου που καθορίζει θεματικούς τομείς στους οποίους θα εργαστεί ο οργανισμός αυτός. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλά πως δεν πρόκειται για ένα πολιετές πρόγραμμα. Ο οργανισμός που είναι εξάρτητος οργανισμός ορίζει κάθε χρόνο το πρόγραμμα εργασίας του. Όμως αυτό το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να καθοριστεί μέσα σε ένα θεματικό πλαίσιο και ακριβώς αυτό είναι ο στόχος αυτής της πρότασης που βλέπετε σήμερα ενώπιόν σας να οριστεί για το έτη 2013 μέχρι και 2017 να οριστούν οι θεματικοί τομεί στους οποίους θα εργαστεί, του οποίου θα ασχοληθεί ο οργανισμό αυτό. Το πολιετέ ε, πλαίσιο των ισχύων ε, εκπνέει στις 31 Δεκάτου 12. Είναι απαραίτητο λοιπόν την 1η Πρώτου 2013 ο οργανισμός να έχει ένα πολιετέ πλαίσιο νέο το οποίο θα έχει οθετηθεί και θα είναι εφαρμοστέο και λειτουργικό. Ποιοι είναι οι θεματικοί τομεί όπου θα εργαστεί λοιπόν αυτό ο οργανισμός. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία ορίζονται στο κανονισμό δημιουργία του οργανισμού. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ο οργανισμός πρέπει να εργαστεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Και οι θεματικοί τομεί βεβαίω θα πρέπει να εντάσσονται στι αρμοδιότητε της Ένωση. Θα πρέπει επίση να αντικατοπτρίζουν τι προτεραιότητε που ορίζονται από την Ένωση, που καθορίζονται μάλλον από την Ένωση. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό είναι ότι οι θεματικοί τομείς θα πρέπει να ορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που υπάρχουν διαθέσιμοι. Πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί όπως το γνωρίζετε είμαστε σε ένα πλαίσιο λιτότητας που όπου πρέπει κανείς να ορίσει πολύ καλά τους θεματικούς τομείς γνωρίζοντας πως ο οργανισμός δεν μπορεί να επεκταθεί σε οποιοδήποτε τομέα. Ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός θα εστιάσει τις δραστηριότητε του και τη συλλογή πληροφοριών για τα θέματα που είναι τα πιο ουσιαστικά για την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη το θέμα των κονδυλίων και αυτό έχει ληφθεί υπόψη από την Κομισιόν. Τελευταίο στοιχείο που είναι επίσης σημαντικό είναι η προστιθέμενη αξία και η μη επικάλυψη. Είναι σαφές πως ο οργανισμός θα πρέπει να εργαστεί σε τομείς που ήδη εξετάζονται από άλλους τομείς, από άλλους οργανισμούς, υπηρεσίες βασικός ρόλος του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι να συλλέγει αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία και υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που εργάζονται σε ορισμένους τέτοιους τομείς. Η Κομισιόν λοιπόν μερίμνησε ώστε οι θεματικοί τομείς να λαμβάνουν υπόψη αυτό το στόχο μη επικάλυψης. Ποιοι είναι οι θεματικοί τομεί λοιπόν, του είδατε στην πρότασή μα. Δεν χρειάζεται να σας του διαβάσω τώρα, να του απαριθμίσω, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αυτοί οι θεματικοί τομείς καλύπτουν την δικαιοσύνη, την ε, κατάσταση θυμάτων ε, δικημάτων, την κοινωνία της ε, πληροφορίας, το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την αστυνομική συνεργασία, την δικαστική συνεργασία, τα δικαιώματα του παιδιού, τις διακρίσεις, τη μετανάστευση, την ένταξη των μεταναστών, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία που είναι μάλιστα μια αναπέτηση που είναι τοποθετημένη μέσα στον κανονισμό που λέει ότι το πολιετές πλαίσιο πάντοτε θα πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας πάντοτε θα πρέπει να εργάζεται για αυτούς τους τομείς αυτός ο οργανισμός. Αυτοί οι τομείς λοιπόν καθορίστηκαν και μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς τα, και κυρίως την κοινωνία των πολιτών και προσπαθήσαμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στο να μπορέσει ο οργανισμός να δουλέψει πάνω στις προτεραιότητες κλειδιά, αλλά προσέχοντας να μην ε, διασκορπιστούν οι δραστηριότητες του οργανισμού που και πάλι, όπως σας είπα, δεδομένου του σημερινού πλαισίου δεν μπορεί να δουλέψει σε όλα τα μέτωπα. Ένα από τα στοιχεία κλειδιά ήταν η συνέχεια, γιατί ο οργανισμός εδώ και κάποια χρόνια έχει αναπτύξει ένα αναγνωρισμένο, μια αναγνωρισμένη τεχνογνωσία όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για διάφορα θέματα. Όλοι γνωρίζουν κάποια προϊόντα του οργανισμού, για παράδειγμα ας πούμε των διακρίσεων, τις μελέτες ε, που είναι σημαντικές ε, ας πούμε στην καταπολέμηση της ε, ε, ομοφιλοφοβίας. Και ε, έτσι μπορέσαμε να διατηρήσουμε ε, πολλά θέματα που υπάρχουν ήδη στο προηγούμενο πολιτές πρόγραμμα, αλλά ένα σημαντικό στοιχείο ήταν η έναρξη ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας, θα έλεγα ότι η μεγάλη καινοτομία σε αυτό το νέο πολιτες πλαίσιο είναι η κάλυψη του πρώην τρίτου πυλώνα, δηλαδή ο τομέας της δικαστικής συνεργασίας σε θέματα ποινικού δικαίου και ε, τα θέματα αστυνομικής συνεργασίας. Είναι τομείς που μέχρι στιγμής δεν καλύπτονταν από το πολιετές πλαίσιο, διότι ο οργανισμός δεν μπορούσε παρά να δουλέψει μέσα στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης. Και πριν από τη συνδίκη της Λαβώνας, ο τρίτος πυλώνας δεν ήταν κομμάτι του κοινοτικού δικαίου. Τώρα όμως ε, που το κοινοτικό δίκαιο είναι το, δικαίωμα ε, το δίκαιο της Ένωσης, μπορούμε να δουλέψουμε και στον τρίτο πυλώνα. Το μόνο εμπόδιο είναι ότι θα πρέπει αυτή, αυτός ο τομής να αναφέρεται και να προβλέπεται στο πολιετές πλαίσιο. Και για αυτό το λόγο, ε, μέσα στο νέο πολιετές πλαίσιο προβλέπεται η ένταξη του θεματικού τομέα της αστυνομικής και της δικαστικής συνεργασίας. Ένα τελευταίο σημείο για την νομική βάση που χρησιμοποιήθηκε. Το πολιετές πλαίσιο βασίζεται στο άρθρο 352 Πράγμα που αιτιολογείται από το γεγονός ότι αντίθετα για τα όσα συνέβαιναν μετά όσα συνέβαιναν για το πρώτο πολιτέ πλαίσιο που βασιζόταν σε μια νομική βάση που προβλεπόταν στον κανονισμό ε, δημιουργίας του οργανισμού μετά από την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που είπε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε παράγωγες βάσεις χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί η νομική βάση δημιουργίας στην οποία βασίστηκε η δημιουργία του οργανισμού, δηλαδή το άρθρο 352, που σημαίνει ότι χρειάζεται έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ ε, δεν ίσχυε κάτι τέτοιο για το πρώτο πολιετές πλαίσιο, όπου δεν υπήρχε αυτή η υποχρέωση. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτή την πρόταση όπως γνωρίζετε, ο Οργανισμός Θεμελιωδών ε, Δικαιωμάτων είναι ένα βασικό εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να δώσει ε, αντικειμενικά και συγκρίσιμα αξιόπιστα στοιχεία για την κατάσταση των ανθρωπίνων των πίνων δικαιωμάτων. Πολύ σημαντικό μέσο εργαλείο για να οριστούν οι τομεί δραστηριότητα του οργανισμού για τα επόμενα χρόνια και η Κομισιόν επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί σα για την συγκεκριμένη πρόταση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you. Ε, ευχαριστούμε. Ο κύριος Μισελ είναι ο πρώτος που έχει το λόγο από τους συναδέλφους που έχουν ζητήσει να παρέμβουν. Μετά από την ε, τροποποίηση του πολιετούς προγράμματος 2007-2012 η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου είχε καταλήξει όπως το είπατε άλλωστε εκπρόσωπε της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι σχετικά με την ε, ποινική και αστυνομική ε, συνεργασία χρειαζόταν να αλλάξει ε, το καθεστώς του γραφείου διαφορετικά θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα κάθε φορά που θέλουμε να ανανεώνουμε το πολιετές πρόγραμμα. Ήθελα όμως να τονίσω και ένα θέμα πιο σημαντικό <clears throat> το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με ε, την συζήτηση που είχαμε πριν από λίγα λεπτά. Δηλαδή ότι το γραφείο αυτό δεν μπορεί να κρίνει μία κατάσταση σε ένα κράτος μέλος αλλά πρέπει να ε, εξετάσει την κατάσταση εγκασίως Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί παραδείγματο χάρη να αποφανθεί στην κατάσταση στην Ουγγαρία οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε τον κανονισμό για να μπορούμε να έχουμε ένα γραφείο γραφείο το οποίο θα είναι ανεξάρτητο, αυτόνομο, με ένα πεδίο ε, δράσεως και ε, ε, δυνατότητα επιβολής ε, Παραδείγματο χάρη ή ε, την περίπτωση παραβιάσεως του άρθρου 7 διότι αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε, κρά... σε περίπτωση ενός κράτος μέλους θεωρούμε ότι είναι κάπως άχρηστο. Δεν μπορεί με να μας δώσει μία εγκάρση αξιολόγηση, αλλά δεν θα έχει παραγματική δυνατότητα δυνατότητα ερεύνης ε, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριε Μισελ. Η κυρία Ιντβελτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βλέπετε ότι ε, τα μισά μέλη που παρίστανται, δηλαδή τέσσερα, συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή. Και είναι κρίμα διότι σήμερα το απόγευμα είχαμε τη συζήτηση και θα ήθελα να πω ότι ε, εξετίμησα τον τρόπο με τον οποίο προεδρεύσατε και δεν συμφωνώ με τον κύριο Μισελ διότι κατόπιν συζητήσεως που είχαμε και τις πολλές συζητήσεις που είχαμε για τις απελάσεις των Ρωμά, ε, για τους ομοφιλοφίλους, όλες τις παραβιάσεις στα κράτη-μέλη, όλα τα θέματα αυτά έπρεπε να είναι στο προσκήνιο και ίσως θα έπρεπε να γίνει μια συζήτηση με περισσότερους παρισταμένους για να συζητήσουμε ε, για την εντολή, για το πλαίσιο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Διότι όταν ε, επισήμως εν ονόματι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ρωτήσαμε πέρσι το, την, το γραφείο να μας πει ποια ήταν η κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη, το γραφείο απλώς ανήθηκε και είπε δεν είναι στην εντολή μας και ούτως ή άλλως δεν έχουμε και τα μέσα. Εφόσον δεν υπάρχει εντολή, τι να τα κάνετε τα μέσα. Λοιπόν, είναι μία <clears throat> απόρριψη, μία άρνηση και πιστεύω ότι το Γραφείο των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει όντως να είναι ουσιαστικό και να μπορεί να επηρεάσει την έκβαση των καταστάσεων και να επιτηρεί ε, την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δίνω λοιπόν τώρα το λόγο πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Απλώς θα ήθελα να διευκρινίσω αυτό το οποίο ελέγχθη και που είναι αρκετά σημαντικό διότι πρέπει να υπάρξει μία διάκριση στη συζήτηση μεταξύ αυτής της προτάσεως που είναι το πλαίσιο που καθορίζει τα θεματικά, τις θεματικές ενότητες και τις άλλες χρήσεις που μπορεί να έχει το γραφείο αν, θέλει να, αν πρέπει να αναλάβει άλλα καθήκοντα, περισσότερους στόχους κτλ. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για τις δραστηριότητες ούτε για τις αρμοδιότητες αλλά αυτό που θα θέλαμε να ξέρουμε είναι αν θα υπάρξει μία αξιολόγηση ο και μπορώ να σας πω ότι θα ξεκινήσει εφέτος ε, η αξιολόγηση του γραφείου από ένα το όργανο το οποίο θα έχει επιλογή βάσει μίας διαδικασίας και θα αξιολογήσει ε, την, ε, το γραφείο αυτό και ε, θα εξεταστεί από ένα διοικητικό συμβούλιο που είναι ανεξάρτητο, δεν εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη και εκεί θα γίνουν ε, ε, συστάσεις στις αρχές του 2013 προς το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για το τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και εκείνη τη στιγμή θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τις αρμοδιότητες, εάν δηλαδή πρέπει να τις προσαρμόσουμε, να δούμε πώς θα τις ε, ε, θα τις εξετάσουμε πράγμα το οποίο δεν είναι εδώ ο στόχος ο στόχος είναι να έχουμε ένα πλαίσιο που χρειάζεται για την 1η Ιανουαρίου του 2013 και να καθορίσουμε τις θεματικές ενότητες και ε, αυτό προβλέπεται στον κανονισμό, δηλαδή να καθοριστούν οι θεματικές ενότητες και να μην αλλάξουμε το σύστημα λειτουργίας του οργανισμού. Ε, όπως γνωρίζουν ε, οι ενδιαφερόμενοι, αυτό είναι σωστό, η συζήτηση ήταν περίπλοκη, ήταν ευρεία, και όταν εφαρμόσαμε τον κανονισμό καταρτήσεως του οργανισμού προβλέφθηκε ένα σύστημα αξιολογήσεως το οποίο θα παρουσιάσει την πρώτη έκθεσή του στις αρχές του 2013 οπότε θα δούμε πώς λειτουργεί και ε, τι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί η λειτουργία της. Θα ήθελα όμως να διευκρινίσω ότι εδώ αναφερόμαστε ε, σε μια διαφορετική πρόταση από τη συζήτηση ε, αυτή η οποία ήταν διαφορετική. Ευχαριστώ. Είμαι βέβαιος ότι για την επόμενη φορά με τους εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές θα έχουμε μία πιο ενεργή συζήτηση στο θέμα αυτό. Τελειώσαμε την εξέταση της ημερησίας διατάξεως, οπότε σας αναφέρω ότι για την επόμενη συνεδρίαση θα συναντηθούμε στις 23 Ιανουαρίου από τις 17 και 15 ως 17 και 45 συντακτική συνάντηση και μετά 25 και 26 Ιανουαρίου θα συνεδριάσουμε τακτικά. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Γεια σας.